Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε αμέσως. Έχουμε αργήσει 12 λεπτά. Θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη It be toast all, but few remarks at the beginning. Mm. Δεν έχω σκοπό να κάνω πρόποση. Κάποιες παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Παρακαλώ κλείστε τα τηλέφωνά σας, αν γίνεται. Και ας πάψουν οι συνομιλίες για να με ακούσετε. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ζητήσω συγγνώμη για αυτή την καθυστέρηση, αλλά ήταν ανάγκη να πάρουμε αυτή την πολύ σημαντική απόφαση στις συνεδρίες των συντονιστών. Υπάρχει ένα ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα για το πακέτο για την καθαρή ενέργεια. Και δυστυχώς καθυστερήσαμε λίγο στη συζήτηση και καθυστερήσαμε και την ψηφοφορία κατά 2-3 εβδομάδες. Παρ' όλα αυτά όμως αποφασίσαμε να τελειώσουμε να ολοκληρωθεί το πακέτο αυτό εντός του 2017. Απλά όχι τον Νοέμβριο, τον Δεκέμβριο. Δεν ήταν εύκολο το να πάρθει απόφαση για το πώς θα προχωρήσουμε από τη μία νομοθετική πρόταση στην επόμενη. Διότι η μία νομοθετική πρόταση μπορεί να επηρεάσει την άλλη. Άρα δεν ήταν εύκολο να ε, καθορίσουμε τη σειρά Εν πάση περιπτώσει, το Νοέμβριο και το Δεκέμβριο αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα υπάρξουν πολλέ ψηφοφορίε για νομοθετικέ προτάσει στην Επιτροπή Ήτρε. Σκληρή δουλειά μα περιμένει. Λοιπόν, και περνάμε στι σημερινέ ψηφοφορίε. Να σα πω ότι θα κάνουμε μία δοκιμαστική ψηφοφορία. Αν δεν γίνει αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Να κάνουμε λοιπόν μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ για να δούμε αν όλα λειτουργούν σωστά. Είστε έτοιμοι να εγκαταλείψετε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πέντε εβδομάδες. Very simple question. Απλό το ερώτημα. Ψηφίστε. Yeah. Has anybody, has everybody, has everybody... Ψήφισαν όλοι. Πέρας ψηφοφορία. Ωραία. Είστε έτοιμοι λοιπόν να αποχωρήσετε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πέντε εβδομάδε. Τέλεια. Γενικό προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το οικονομικό έτο 2018, όλα τα τμήματα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τροπολογία 177. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Να ελέγξουμε. Να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 184 υπέρ κατά ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα για την 184. Ένας πλεονάζων από το ΕΛΚ. Πέρασε της Εγκρίνεται. 1.57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 40 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 175 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 69 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 176 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 172 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 140 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 159 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 92 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 93 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 94 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 95 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 97 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 151 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 185 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 158 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 152 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ...173 υπέρ... ...κατά... ...αποχές... ...απορρίπτεται... ...127 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 174 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται, 128 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τώρα, ψηφοφορία unblock, 1 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Block vote 2. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Είμαστε στη σελίδα 12. 160. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 167. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 198. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 179. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 180. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 166 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 189 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 191 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 190 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 202 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 206 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 186 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 187 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 188 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 192 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 193 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 194 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 199 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 201 υπέρ 201 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 203 υπέρ κατά αποχές Καλύτερα να πείσουμε ηλεκτρονικά. Ας ελέγξουμε λοιπόν Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 203. Ένας πλεονάζων από το ΕΛΚ. Πέρα στις ψηφοφορίες. Εγκρίνεται. 205 υπέρ, κατά. Μα δεν ψηφίζετε. Ξανά. Πάμε. 205 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα ήταν σαφές. 200 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 182 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 183 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 195 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 163 υπέρ, κατά, επί της διαδικασίας, κύριε Τούρνες. υπάρχουν δύο πολιτικά προγράμματα. Εδώ, αν μάλιστα διαβάσετε τον τίτλο, είναι και τον δύο, είναι πολύ παρόμοια. Μα αυτό δεν είναι διαδικαστικό, λέει ο Πρόεδρος, έχουμε συζητήσει το θέμα αυτό. δεν έχουμε τώρα αυτή τη δυνατότητα να μιλήσουμε επί της ουσίας. Ξανά, 163 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 164 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 170 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 161 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 207 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 204 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τέλος εφορία. Γιατί ψηφίζουμε μόνο γραμμές του προπολογισμού. Τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει ούτε ψήφισμα, ούτε άλλη απόφαση που λαμβάνεται. Ψηφίσαμε λοιπόν όλες τις γραμμές του προπολογισμού και θα αποσταλεί τώρα η, ε, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας μας στην Επιτροπή Προπολογισμού. Τώρα λοιπόν περνάμε σε ένα πολύ πιο δύσκολο θέμα. Θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη γιατί θα αναγκαστώ να σας ε, ζητήσω να, το, να ελέγξετε το αποτέλεσμα. Γιατί οι πολιτικές ομάδες είναι διχασμένες. Δεν αρκεί εγώ να βλέπω τι ψηφίζουν οι συντονιστές. Γιατί εσωτερικά οι πολιτικές ομάδες είναι διχασμένες, δεν έχουν κοινή στάση. Οπότε φαντάζομαι ότι θα γίνουν πάρα πολλές ηλεκτρονικές ψηφοφορίες σε αυτή την περίπτωση. Ας ξεκινήσουμε θέλω απλώς να εξασφαλίσω πως έχει αποσυρθεί η τροπολογία 234. Ευχαριστούμε. Ωραία, ας ξεκινήσουμε λοιπόν εκατόν 29 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Για τη συμβαστική 1. Συμβαστική 0. Υπέρ, κατά, αποχές, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Συμβαστική 0. Πέρας. Υπεράριθμοι. Ένας πλεονάζουν από το ΕΛΚ. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται η συμβαστική τροπολογία 0. 130 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 131 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τώρα θα ψηφίσουμε από κοινού. Συμβαστική 1, συμβαστική 2, συμβαστική 2α, συμβαστική 3, συμβαστική 3α. Τρεις συμβαστικές. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 1α. We, we, we voted. It was, it was rejected. I wanted to check. Uh, do you want to, to check it? Θέλετε να το ελέγξουμε. Όχι, κανείς δεν ζήτησε να γίνει έλεγχος. Βάση περιπτώσει. Λοιπόν, θα, θα ε, ψηφίσουμε τώρα για αυτές τις ε, πέντε συμβαστικές. Πέρας της προφορίας. απορρίπτεται. Συμβαστική 1α υπέρ, κατά, αποχές, ας το ελέγξουμε καλύτερα. Πέρας της Πέρας Ξαναλέω. Εγκρίνεται. Εγκρίνεται η συμβαστική Τροπολογία 1α. 1 to 140. 140. Page 6. We gone, it was accepted. We go to page 6. Αφού εγκρίθηκε πάμε στη σελίδα 6. Ε, συμβαστική 140. Σελίδα 6. 140. Υπέρ, κατά, Ας πάμε κατευθείαν σε ηλεκτρονική ψηφοφορία γιατί δεν ξέρω πώς ψηφίζετε. Μιλάμε για την τροπολογία 140. τη ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 152 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 153 υπέρ, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για την 152. Ας το ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος της ψηφοφορίας. ΕΛΚ είστε υπεράριθμοι. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Απορρίπτεται. 153. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές, καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ για την τροπολογία 154. Τέλος της προφορίας. Πάλι ένας παραπάνω από το ΕΛΚ. Θα βγάλω εγώ την κάρτα μου στο τέλος. Απορρίπτεται. 151 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 155 υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 4 υπέρ, κατά, νομίζω ότι εγκρίνεται, αλλά καλύτερα να ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Α το ελέγξουμε, ψηφίστε παρακαλώ. I close the vote. Compromise 4. Accepted. Συμβαστική 4. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 165. Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 166. 173 από κοινού υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 168 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 169 υπέρ κατά, να το δούμε ηλεκτρονικά. 169. Λίγοι. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 171 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 172 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 178 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 179 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 180 υπέρ κατά αποχές α, να το δούμε και ηλεκτρονικά 180 180 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 181 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, συμβαστική 7 ε, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 184 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 185 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 186 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 187 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές Απορρίπτεται. Ωραία. Ελεκτρονικά, λοιπόν τη συμβιβαστική 8. Λίγη ψηφοφορία. Απορρίπτεται. Και μετά έχουμε τέσσερις τροπολογίες μαζί. Μία 88, μία 89. Συγγνώμη, 188, 189, 190 και 191. Μαζί. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 192 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και μετά, πάμε στην 193, που είμαστε υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 194 και 195 μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 196 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 197 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 198 υπέρ, αποχές, κατά, απορρίπτεται. 199 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 200 υπέρ, κατά, για να δούμε τη 200 ηλεκτρονικά. 200, ε, πέρας ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 201 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 202 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 203 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονικά τη συμβαστική 10 πέρας πληροφορίας εγκρίνεται συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται την 11 ηλεκτρονικά Συμβιβαστική 11. Ηλεκτρονικά. Πέρας. Απορρίπτεται. 216 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 209 υπέρ. Κατά για να τη δούμε ηλεκτρονικά. 209. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 207 υπέρ. Συγγνώμη. 217 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 213 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 214 υπέρ, κατά, συγγνώμη, 224 υπέρ, κατά. Α, έχει, έχει αποσυρθεί. 233-234 έχουν απορριφθεί. 2.48 υπέρ. Κατά. Για να θα δούμε. 248 ηλεκτρονικά. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 16 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.45 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.46 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.47 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.49 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.50 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 2.51 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 2.52 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.53 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 2.54 υπέρ, κατά. Για να το δούμε ηλεκτρονικά. 2.54 ηλεκτρονικά. Πέρας πληροφορίας. Απορρίπτεται. 2.55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.58 μαζί με τη 2.59 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά για να το δούμε ηλεκτρονικά. Ηλεκτρονικά λοιπόν, στην 13, τροπολογία 13, πέραση ψηφοφορίας, απορρίπτεται. 14 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 15 υπέρ, κατά. Για να το δούμε ηλεκτρονικά λοιπόν, την 15, για να Ελέγξουμε τη 15. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 17α συμβαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Θέλετε να δούμε ηλεκτρονικά τη 17α. Μπορεί να είναι πραγματικά κοντά τα νούμερα. Λοιπόν, συμβιβαστική 17. Πρώτα απ' όλα ηλεκτρονικός έλεγχος της 17. Ξεκινάμε λοιπόν με τη 17. Μία πίσω ψηφίζουμε, τη 17. Συμβιβαστική 17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 17α. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική 18 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται με την ίδια πλειοψηφία. 18α συμβιβαστική υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, η 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Η 26 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19α υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Συμβιβαστική 20 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21α υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 22α υπέρ 22α κατά αποχές εγκρίνεται. 22α είναι δεκτή. 22 απορρίφθη. Η τροπολογία 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπεται. 47 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτε. συμβαστική 26 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 28 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 29 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 55 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτε. 56 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται η 57 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 58 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 59 υπέρ κατά για να το δούμε την 59 παρακαλώ ηλεκτρονικά πέρας Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική. Α, συγγνώμη. 62 63 μαζί. 62 και 63 μαζί. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 64 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 65-66 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68, 69 και 70 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 72 υπέρ κατά αποχές αποδεκτή εγκρίνεται λοιπόν 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 74, 75 και 76, 74 και 75 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 76 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 79 και 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 81 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά για να δούμε την 82 ηλεκτρονικά παρακαλώ πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 83 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 91. Φτάνουμε λοιπόν στην 91. 91 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 36 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Και μετά τέσσερις τροπολογίες μαζί. 102, 103, 104 και 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 123 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 124 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές την 127 ηλεκτρονικά παρακαλώ 127 πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Και 128 υπέρ, κατά, αποχές. Για να δούμε και την 128 ηλεκτρονικά παρακαλώ. 128 ηλεκτρονικά. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Και τώρα τελική ψηφοφορία ονομαστικά. I open the vote. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. 39-18. Έξι εποχές. Συγχαρητήρια. Δεν ήταν εύκολη η δουλειά μας. Συγχαρητήρια στον εισηγητή. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφοι. Ήσασταν πάρα πολύ υπομονητικοί.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

για τον ወγγέλη το πρόβλημα Uh, Επιτρέψτε μου, ενώ προετοιμαζόμαστε για το επόμενο σημείο, να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τους διερμηνείς μας. Ευχαριστώ όλους σας, ελπίζω που με ακούτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, λέει στα πολωνικά ο Πρόεδρος, τους διερμηνείς τους άντρες και τις γυναίκες που εργάστηκαν χθες 15 λεπτά παραπάνω. Ήταν πολύ ζωντανή ζωή συζήτηση και χάρη στους διερμηνείς ε, μπορέσαμε να συνεχίσουμε διότι τα μέλη μας δεν ήξεραν ποια ε, γλώσσα να χρησιμοποιήσουν για κοινή συνεννόηση. Ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ που εργαστήκατε χθε ένα τέταρτο περισσότερο. Δεν συμβαίνει αυτό πάρα πολύ συχνά, αλλά η συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή. Ξέρω ότι οι ίδιες ομάδες εργάζονται σήμερα, οπότε σας ευχαριστώ για αυτό. Πάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης στην Επιτροπή Ήτρε μετά την ψηφοφορία προετοιμασία για αντιμετώπιση κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, ο συνάδελφος Φλάβιο Ζανονάτο είναι ο εισηγητής. Το θέμα αυτό είναι ένα κομμάτι του πακέτου για την καθαρή ενέργεια και συνδέεται με την οδηγία για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τον κανονισμό Acer. Ίσως το γνωρίζετε, θα ψηφίσουμε το Δεκέμβριο την όλη δεσμομέτρων για την ηλεκτρική ενέργεια. Θα ψηφίσουμε το Δεκέμβριο, όχι τον Νοέμβριο. Ήταν πρωινή απόφαση αυτή. Προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι κάπως αργότερα, διότι ψηφίζουμε και αργότερα, 13 Σεπτεμβρίου. αργότερα, όχι αρχές Σεπτεμβρίου, αλλά 13 Σεπτεμβρίου. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσπαθεί να εξασφαλίσει ότι όλα τα κράτη-μέλη θα θεσπίσουν κατάλληλα εργαλεία για να είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν η αδίποτε κρίση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ετοιμότητα λοιπόν για αντιμετώπιση κρίσεων. Κύριε Ζανονάτο, αγαπητέ συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Τώρα η διαχείριση για την αντιμετώπιση των κινδύνων στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας είναι θέμα σχεδόν αποκλειστικά εθνικής ε, αρμοδιότητας. Σύμφωνα το άρθρο 194 των συνθήκων, η ενεργειακή πολιτική της Ενώσεως δεν έχει εργαλεία για να εγγύεται την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια, μέσω μηχανισμών προλήψεως, προετοιμασίας, διαχείρισης, αξιολόγησης, εκ των υστέρων των διαφόρων υποθέσεων για κρίση στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Λοιπόν, εντάσσεται στην αξιολόγηση των διαθεσίμων υποδομών αντιμετώπιση των κρίσεων με αποτέλεσμα ότι είναι ελεύθερα τα κράτη-μέλη να καθορίσουν τις δράσεις και τα μέτρα τα για να διαχειριστούν και οι δυνατόν να ξεπεραστούν οι κρίσεις του συστήματος. Όμως σε μια αγορά ενεργειακή που σταδιακά ολοκληρώνεται, τα εθνικά μέτρα και διορθώσεις ε, κινδυνεύουν να είναι αναποτελεσματικά μέτρα. Υποδειγματικό η υπόθεση είναι τον περασμένο Ιανουάριο η κρίση που ξέσπασε στην νοτιοδυτική Ευρώπη. Υπάρχει νομοθετικό κενό και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε έναν κανονισμό που έχει σαν στόχο να αυξήσει τη συνεργασία μεταξύ κρατών μελών στον αφορά την πρόληψη προετοιμασία και διαχείριση ενεργειακών κρίσεων. Είναι ένα κείμενο που στη δομή και διάθρωσή του γενικώ θεωρώ ότι είναι κάτι θετικό, το βλέπω θετικά το κείμενο. Τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την αντιμετώπιση οικονομικών ζημιών και των τιμολογικών συνεπιών και των ε, επικινδύνων συνεπιών για την παροχή των ουσιαστικών και βασικών ε, παροχών ηλεκτρικής ενέργειας ε, τα προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν σε περιοχές των κρατών μελών. Ε, έχω τρία σημεία που θέλω να φέρω όσον αφορά την πρότασή μου. Συνεργασία και αλληλεγγύη είναι το πρώτο σημείο για να εξασφαλίσουμε σωστές ανταλλαγές πληροφοριών για την κρίση την, στον τομέα ηλεκτρικής ενέργεια πρέπει να είναι προσβάσιμα όλα τα στοιχεία όσον αφορά περιφερειακά σχέδια αντιμετωπίσεως του κινδύνου. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συντονίζονται μια μεθοδολογία περιφερειακή κοινή που θα πρέπει να εφαρμόσει. Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να υπενθυμίσουμε κιόλα ότι τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε ξεχωριστές αξιολογήσεις και να δουν πώς βραχυπρόθεσμα ποια υπάρχει και υπάρχει για να μπορούν να ανταποκρίνονται στις απαιτήσει και στα χαρακτηριστικά τα αντίστοιχα. Τα μεθοδολογικά κριτήρια κοινά είναι ένα στοιχείο απαραίτητο για να ενισχυθεί η αρχή της συνεργασίας κυρίως σε τεχνικό επίπεδο μεταξύ των TSOs και πιστεύω ότι μετά όλες τις εμπειρίες κατά τη διάρκεια της ενοποίησης των διαφόρων περιφερειακών συντονιστών για την ασφάλεια του RSC είναι μια προσέγγιση προς αυτή την κατεύθυνση. Όσον αφορά την πολιτική πτυχή για τη συνεργασία και την αλληλεγγύη μεταξύ 100 μελών, το σχέδιο τη εκθέσεω επιβεβαιώνει την αρχή τη αμοιβαία αρρωγή που προτείνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και περιορίζεται έτσι το πεδίο των παρεκκλήσεων όσον αφορά το, λόγω των εμποδίων ε, τεχνικής φύσεως. Τροπολογία 19. Θα πρέπει λοιπόν να οριμάσει το όλο ηλεκτρικό σύστημα, να υπάρχει η αυξανόμενη διασύνδεση μεταξύ των περιφερειών περιφερειών τη Ευρώπη και λαμβάνοντας υπόψη την εξέλιξη των αγορών και σε πολύ βραχυπρόθεσμη περίοδο, δεν μπορεί να είναι απομονωμένε διάφορες περιοχές ενεργειακά. Κυρίω οι χώρε που κινηθούν προς αντίθετη κατεύθυνση. Γι' αυτό μηχανισμοί αντισταθμιση μεταξύ κρατών μελών που αντάλλαξαν ενέργεια λόγω ηλεκτρική κρίσεως θα πρέπει να καθορίζονται ανάντι σε περίπτωση κρίσεως και όποτε είναι δυνατόν ή τουλάχιστον στην αρχική φάση που ξεσπάει η κρίση λήψη σχημάτων ε, ε, αντιστάθμισης θα είναι πολύ πιο δύσκολο να εγγυηθούμε την εφαρμογή της αρχής αμοιβαίας αρρωγής. Σημείο 2 προδιαγραφές της αγοράς ε, και αποθεματοποίηση. Μια κρίση στον τομέα ηλεκτρικής ενεργείας δεν μπορεί να είναι άλοθη για προσφυγή σε μέτρα βελτιστοποίησης της αγοράς. Και από αυτήν την οπτική γωνία οι προδιαγραφές όχι της αγοράς θα πρέπει να θεωρηθούν αποδεκτές μόνο όταν οι κανόνες αγοράς κινδυνεύουν να επιδεινώσουν μια κατάσταση κρίσεως. Και αυτήν την τροπολογία 20 όσον αφορά την το περιεχόμενο των σχεδίων και την αποκάλυψη των σχεδίων πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ε, μεταχείριση των ευαισθητών στοιχείων, κυρίως στα περιεχόμενα των σχεδίων που θα μπορούσαν να εκθέσουν τα επιχειρησιακά ε, σχέδια σε επιθέσεις τρίτων τρομοκρατών ή ε, διαφόρων κακοποιών στοιχείων. Και αυτό είναι στην τροπολογία 16. Τελευταίο σημείο διακυβέρνηση. Ε, μια ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο άρθρο 12 που αναφέρεται δυνατότητα διαφωνίας μεταξύ των αρμοδίων αρχών και τη δυνατότητα που έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητήσει από την Acer να διευκολύνει μια συμφωνία κατόπιν διαβούλευση με του αρμοδίου φορεί. Πιστεύω ότι αυτή η διατύπωση δεν είναι αρκετά σαφή, κυρίω σε σχέση με τα διάφορα καθήκοντα για τη λήψη αποφάσεων. Για να μην υπάρχουν αμφιβολίε, προτείνω την τροπολογία 17 για να προσφύγουμε στο μηχανισμό συνεργασία ε, και σε συντονισμό με τον κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού φυσικού αερίου ο μηχανισμό συνεργασία διευκολύνει και διαθρώνει τη σύναψη μια συμφωνία όσον αφορά τα περιφερειακά μέτρα. Αλλά η απόφαση η τελική όσον αφορά τα περιφερειακά μέτρα παραμένει στα χέρια των αρμοδίων αρχών των κρατών μελών που τα αφορά. Επιπλέον πιστεύω ότι η διακυβέρνηση σημαίνει επίσης πλήρη συμμετοχή του διαχειριστού του συστήματο μετάδοση ενέργεια και των διαχειριστών του συστήματων διανομή για τον εντοπισμό και την προετοιμασία και τη διαχείριση και τον έλεγχο και τη διαδικασία αξιολογήσεως των υστέρων της κρίσεως. Από την άλλη πλευρά, αυτοί οι φορείς της αγοράς είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την αξιοπιστία της λειτουργίας του συστήματος. Τέλος, κλείνοντας, προτείνω και πιο λειτουργική και οθολογική στάθμιση του χρόνου εκτέλεσης των διαφόρων φάσεων και ταυτοχρόνως πιστεύω ότι εκ των υστέρων αξιολόγηση μπορεί και θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει την ανάλυση του τρόπου με τον οποίο το δίκτυο θα μπορούσε να αναπτυχθεί ούτως ώστε να αντιμετωπίζει καλύτερα τις συνέπειες κρίσεως που εντοπίζονται. Εάν αυτή η πρόταση του κανονισμού ε, είναι νόμος, όπως το θέμα της διαχειρίσεως των κινδύνων που καλύπτει το, τις φάσεις πρόληψης αξιολόγησης εκ των υστέρων των κρίσεων περιφερειακών στην Ευρώπη Ταυτόχρονα χρειάζεται σε αυτές τις κρίσεις, σε αυτές τις κρίσεις να έχουμε τη μεγίστη συνεισφορά των πληροφοριών που μπορούν να επεξεργαστούν. Ούτω ώστε να υπάρχει ασχεδιασμό μέσω μακροπρόθεσμο όσον αφορά τι απαιτήσει ανάπτυξη ε, του μελλοντικού δικτύου ηλεκτρική ενεργεία και υπό το φω ε, τη κρίσεω. Από αυτήν την άποψη. Είμαι ικανοποιημένο που άκουσα να ακούσω τη συνεισφορά των συναδέλφων δέκτο ε, καλύπτει μεγάλα κενά υπό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αλλά σε κάποιες λεπτομέρειες μπορεί να βελτιωθεί αυτό που ανέφερα. Χρειάζεται συνεργασία, αλληλεγγύη, άνοιγμα των αγορών και ταυτόχρονα πρέπει να προστατεύονται τα συστήματα από κινδύνους επίθεσης. Και όσον αφορά τη διακυβέρνηση, χρειάζεται σαφέστερο ορισμό. Δεν θέλω να συνεχίσω, διότι θέλω να ολοκληρώσω και θέλω να ευχαριστήσω όλου για τι ε, συνεισφορέ του που θα ακούσω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ 8 λεπτά είχατε στο, συνολικά. Στο, στο τέλος θα σας παρακαλέσω. Μιλάνε και οι δύο μιλτές μαζί, μπα τους καταλάβουν δυστυχώς. Λέω, ο Πρόεδρος. Μισό λεπτό θα σας δώσω στο τέλος για να συνοψίσετε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τις πολύ ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις σας και για την έκθεσή σας φυσικά. Ο συνάδελφος Νίντερμαερ εκ μέρους του ΕΛΚ, Σκιώδης. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πολύ σημαντική η έκθεση αυτή, όχι μόνο γιατί εντάσσεται εντό τη δέσμη μέτρων, αλλά γιατί είναι και μια λογική συνέπεια των αλλαγών που συμβαίνουν στην ηλεκτρική, στον τομέα τη ηλεκτρική ενέργεια ε, και τις αλλαγές ε, στην, ε, στη δομή της αγοράς. Ταυτόχρονα το μερίδιο της ηλεκτρικής ενέργειας στην συνολική ποσότητα ενέργειας που καταναλώνεται αυξάνεται οι εθνικές αγορές δεν είναι επαρκώς διασυνδεδεμένες. Γι' αυτό και ε, πρέπει να εξεταστεί ε, η δραστηριότητα των TSO. Οι κρίσεις μπορούν να είναι εγγενείς, ε, εθνικές ή και ε, εισαγόμενες, αλλά το ίδιο ισχύει και για τις λύσεις στα προβλήματα. Γι' αυτό και είναι σημαντικό να, το γεγονός ότι έχουμε αυτή την πρόταση, που είναι πολύ έγκαιρη. Όπως βλέπω από τις ε, συναντήσεις των σκιωδών η πρόταση αυτή χαίρει της εκτίμησης των περισσότερων, γι' αυτό και νομίζω ότι μπορούμε να ε, καταλήξουμε σε μια ολοκληρωμένη θέση του Κοινοβουλίου, αλλά βεβαίως θα ακούσω και τις απόψεις των άλλων σκιωδών. Παρ' όλα αυτά, θέλω από τώρα να ε, ευχαριστήσω τον εισηγητή για, μια πολύ την, για την πολύ ισορροπημένη του έκθεση. Να επισημάνω τους εξής τομείς θα πρέπει στη διαδικασία αυτή να ε, συμπεριλαμβάνονται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς. TSO, DSO και παραγωγή. Επίσης, πρέπει να τονιστεί η προσέγγιση που θα βασίζεται στην αγορά. Θα πρέπει ε, να εξαντλούνται όλες οι δυνατότητες και στη συνέχεια να λαμβάνονται μέτρα ε, τα οποία όμως δεν θα διαστρεβλώνουν την ε, εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τον ανταγωνισμό. Είναι ευρύτερο το θέμα αυτό όμως, διότι το βασικό σημείο του πακέτου είναι ότι ε, θα πρέπει να αρθούν εμπόδια και στρεβλώσεις αγοράς προκειμένου η τροφοδοσία να, γίνεται, να γίνει φθηνότερη και πιο αξιόπιστη. Τρίτον, Πρέπει να εξασφαλίσουμε ε, την εμπιστευτικότητα των ε, ε, πληροφοριών, ιδίως των πληροφοριών που μπορούν να αξιοποιηθούν από κακόβουλες επιθέσεις. Ξέρω ότι ήδη καλύπτεται το θέμα αυτό στην έκθεση, αλλά πρέπει νομίζω να το αναπτύξουμε περαιτέρω. Και τέλος, ε, νομίζω ότι η συνεργασία ε, θα πρέπει να υπερβαίνει τα όρια της ε, ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμπεριλάβει και τις χώρες της ενεργειακής κοινότητας. Ε, η έκθεση λοιπόν αφορά τη διαχείριση των κινδύνων. Πρέπει να βελτιωθούμε και για να γίνει αυτό πρέπει να ενθαρρύνουμε την περιφερειακή συνεργασία και νομίζω ότι αυτό είναι ο σωστός δρόμος. Αλλά αυτό δεν είναι μόνο σημαντικό για την ετοιμότητα. Νομίζω ότι γενικά η περιφερειακή συνεργασία θα πρέπει να βελτιστοποιήσει την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και όχι μόνο να αντιμετωπίζει τους κινδύνους blackout, αλλά να αξιοποιείται και ε, ε, για την, καλύτερη εξοικονόμηση κόστους και πόρων. Κάτι που θα αποβεί ε, προς όφελος τόσο των πολιτών όσο και των επιχειρήσεων. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάλλας, εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Ναι, εκπροσωπώ τον σκιώδη μας. την σκιώδη μα, που ζητά συγγνώμη που δεν βρίσκεται εδώ σήμερα. Χαιρετίζει το σχέδιο έκθεση του εισηγητή για τους νέους κανόνες για την ετοιμότητα στον ε, τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, την βελτιωμένη συνεργασία, την ενισχυμένη διαφάνεια και την ανταλλαγή πληροφοριών που είναι σημαντικά στοιχεία όχι μόνο στην αντιμετώπιση κρίσεων αλλά και προϋποθέσεις για την οικοδόμηση μιας ανθεκτικής ένωσης ο εισηγητής προτείνει κάποιες σημαντικές διατάξεις για την ενίσχυση της πρότασης της Κομισιόν, ιδίως όσον αφορά την προστασία της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών έναντι κακόβουλων επιθέσεων και την εμπλοκή όλων των φορέων στη διαδικασία. Επίσης, η σκιώδης μας χαιρετίζει την προσπάθεια του εισηγητή να εξασφαλιστεί ε, μεγαλύτερη εναρμόνιση και ε, ευθυγράμμιση. Για να ε, ενισχυθεί ακόμη περισσότερο η πρόταση, η ισχυώδης μας σκοπεύει να υποβάλει προτάσεις που θα αποσαφηνίζουν τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των εθνικών αρχών τις, ε, ε, τα μέτρα αλληλεγγύης και τα ε, ζητήματα που σχετίζονται με τις κρίσιμες υποδομές και τα σχετικά δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση χρειάζεται να αναφερθεί και να, και να καταρτιστεί μάλλον ένα πρόγραμμα ε, αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων και κρίσεων. Και όπως ε, είπα και στην αρχή, η σκιώδης είναι στη διάθεση όλων των υπολείπων σκιωδών για μια ε, καλή συνεργασία. Ο κύριος Τούρμς. Θα συνοψίσω λίγο λέγοντας πως καταρχήν ότι η Γαλλία έφτασε πολύ κοντά σε ένα τεράστιο blackout. Γιατί? γιατί είχαμε η ηλεκτρική θέρμανση συν ε, μη ε, αξιόπιστη πυρηνική ενέργεια οδήγησε σε σχεδόν κρίση χωρίς να υπάρχει κάποιο προληπτικό σχέδιο. Και μόνο την τελευταία στιγμή κατάφεραν να συμφωνήσουν οι TSO και να, οι και να σώσουν τη Γαλλία από, την, ε, τον blackout. Και νομίζω είναι χειρότερη κατάσταση από ό,τι είχε συμβεί τότε με Βουλγαρία, Ρουμανία, Ελλάδα. Αυτή ήταν μια μικρή κρίση και στη Γαλλία δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν τίποτα, έκλεισαν τα σύνορα και επειδή ήταν μια καθαρά εθνική προσέγγιση χρειάστηκε να κλείσουν ε, και τα, ε, τα εθνικά δίκτυα γιατί δεν υπήρξε εσωτερικός συντονισμός. Για να εξηγήσω λοιπόν, το 2006 είχαμε ένα τεράστιο blackout στην Ευρώπη το οποίο προκάλεσε μη συντονισμός ε, ε γερμανικής εταιρείας που κάπου δεν μπόρεσε να περάσει ένα καράβι και εκατομμύρια πελάτες εκτός Γερμανίας έμειναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και ακόμα δεν έχουν πληρωθεί αυτοί οι άνθρωποι κάποια αποζημίωση. Οπότε δεν έχουμε λυγή, δεν έχουμε αποζημιώσεις και δεν έχουμε και προληπτικά ε, σχέδια. Τι να σας πω κύριε Σανωνάτο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσέγγισή σας, κυρίως για το κομμάτι που επιμένει στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας και κάτι το οποίο βρίσκω αρκετά παράξενο στο σχεδιασμό της αγοράς, ο εισηγητής μειώνει τα επίπεδα περιφερειακού συντονισμού διαγράφοντας κάποια σκέλη αυτού του ε, ε, προληπτικού σχεδίου αντιμετώπισης ε, κινδύνων. Οπότε αυτό πρέπει να το συζητήσουμε. Και νομίζω ότι αυτή η αποδυνάμωση της περιφερειακής ε, συνεργασίας θα πρέπει να αντιστραφεί. Αντίθετα, θα πρέπει να πιέσουμε έτσι ώστε να έχουμε μεγαλύτερη συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κωνσταντάμς και παρακαλώ, θα ήθελα εκ μέρους του κύριου Φόξ, που είναι ο σκιώδης μας, να ε, διαβάσω ένα ε, σημείωμα. Η ομάδα μου χαιρετίζει και την πρόταση και το σχέδιο έκθεσης του εισηγητή που θα κάνει πιο ανθεκτική την, το κλάδο του της ηλεκτρικής ενέργειας. η κυβερνοτρομοκρατία η οποία αυξάνεται δημιουργεί μεγαλύτερη πτυτικότητα και οι, οι πιέσει οι γεωπολιτικές σημαίνουν ότι μπορεί να έχουμε πιο σύντομα και είναι πιο πιθανό να έχουμε μια κρίση στο ηλεκτρικό ρεύμα. Άρα λοιπόν η κοινή μεθοδολογία σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να αντιμετωπίζουμε ενδεχόμενες κρίσεις και η ε, τα σχέδια εθνικής και περιφερειακής αντιμετώπισης, το πλαίσιο αξιολόγησης και επιτήρηση είναι όλα πολύ σημαντικά στοιχεία. Όμως λυπάμαι πως το χρονο... Ε, φοβάμαι πως το χρονοδιάγραμμα με τους δύο μήνες για διαβούλευση της μεθοδολογίας και έξι ε, μήνες μετά για την αξιολόγηση κινδύνου και οι δύο μήνες για το εντυπισμό των εθνικών σχεδίων είναι υπερβολικά αυστηρά. Στο άρθρο 5 και 8 θα υποβάλω τροπολογίες για αυστηρότερη ορολογία για τους διαχειριστές ε, συστημάτων διανομής και μεταφοράς, γιατί είναι απόλυτα απαραίτητο να συνεργάζονται για να έχουμε ασφάλεια ανεφοδιασμού. Συμφωνώ με τη διάταξη υπέρ ενό μηχανισμού που θα βασίζεται στις ανάγκες αγοράς και μηχανισμοί εκτός αγοράς θα πρέπει να αποτελούν ε, τελευταίο καταφύγιο και να τεκμηριώνεται η ανάγκη χρήση τους επαρκώς για την αποζημίωση νομίζω ότι θα πρέπει αυτά να οριστούν εκ των προτέρων και να μην επιβάλλονται ε, αυθαιρέτως. Χαιρόμαστε για το γεγονός ότι εδώ έχουμε πλέον το απόρριτο των ευαίσθητων πληροφοριών. Το άρθρο 16 τέλος, εδώ πρέπει να γίνει η επιτουσιολογική μελέτη ε, για το τι θα, πώς θα επηρεαστούν ε, μετά την κρίση όλοι οι εμπλεκόμενοι όπως επίσης και οι παραγωγικές μονάδες. Και με μεγάλη χαρά θα συνεργαστώ με όλους για το συγκεκριμένο θέμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος ομιλητής, ο κύριος Μπενίτο Σιλουάγα. Εμείς πιστεύουμε πως αυτή η έκθεση θα πρέπει να έχει ως στόχο να αναγνωρίσει πως τα μέτρα είναι αρκετά και πως χρειάζεται αυτορύθμιση του κλάδου. Διαφορετικά μπορεί να έχουμε προβλήματα με τον ανεφοδιασμό. Όταν μιλάμε για ασφάλεια. Θα πρέπει να εγκαταλείψουμε αυτό το μάντρα της αγοράς που θα τα λύσει όλα και να δώσουμε μια προτεραιότητα στη δημιουργία κανόνων οι οποίοι θα βασίζονται στην αμοιβαία συνεργασία και στην αλληλεγγύη μεταξύ κρατών μελών. Παρ' όλα αυτά θα πρέπει να λάβουμε επίσης υπόψη το πόσο προσεκτικά θα πρέπει ε, να αναλάβει το δίκτυο ενεργειακών επιχειρήσεων στα πλαίσια της αυτορύθμισης γιατί δεν πιστεύουμε πως είναι η πιο κατάλληλη οντότητα για να, συστή, για να ε, συγγράψει αυτά τα σχέδια έκτακτης ανάγκης που θα πρέπει να συνταχθούν από ε, τον οργανισμό που εκπροσωπεί τα κοινά συμφέροντα στην Ευρώπη. Είναι ολιγοπολιστική εδώ η αγορά και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί με την συγκέντρωση πληροφοριών. Γιατί θα πρέπει να φροντίσουμε αυτό να μην έχει αρνητικέ συνέπειες για την ασφάλεια, άρα χρειαζόμαστε τη μέγιστη δυνατόν διαφάνεια. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Ο κύριος Κόκιτσεκ, αντιπρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να κάνω και εγώ κάποιες παρατηρήσεις. Έτσι ώστε να είναι πιο ζωντανή η συζήτηση για την ηλεκτρική ενέργεια, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε δύο είδου κινδύνους. Καταρχήν τα blackout και το δεύτερο είναι να έχουμε υπερβολικά μεγάλη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος, ηλεκτρικής ενέργειας, ε, να μπαίνει υπερβολικά πολύ ε, ηλεκτρική ενέργεια στο σύστημα. Και τα δύο αποτελούν κίνδυνο και κάποιες ΑΠΕ δεν μπορούν να ρυθμίσουν αυτές τις εισρωές και η μοναδική δυνατότητα είναι να κατεβάσουμε το διακόπτη ορισμένες φορές. Και όπως και οι συνάδελφοι από τους πράσινου, ε, πράσινους είπαν πολύ σωστά, είναι ακριβώς αυτές οι πηγές οι οποίες διακυβεύουν τη σταθερότητα του συστήματος, γιατί εδώ δεν μπορούμε να το ρυθμίσουμε. Και γι' αυτό έχουμε αυτή τη στιγμή τους σταθμούς διαχωρισμού στα, στα πολωνικά σύνορα, όπως επίσης και στα τσεχικά σύνορα, γιατί οι Γερμανοί προμηθευτές δεν κάνουν αυτή τη ρύθμιση και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να το συμπεριλάβουμε και στην έκθεση να πούμε πως υπάρχει ένα μεγάλος κίνδυνος για, την, ε, για τα αποθέματα και τον εφοδιασμό σε ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι μόνο το downtime που είναι κίνδυνος δεν είναι μόνο η έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας αλλά είναι και η υπερβολική ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να μας δυσκολέψει και αυτή η σταθμή διαχωρισμού μπορεί από μόνοι τους να, να προκαλέσουν blackout. Η καλύτερη δυνατότητα είναι όχι περισσότερη αγορά, αλλά περισσότερη συνεργασία. Η TSO των 16, και εδώ συμπεριλαμβάνω την Ουγγαρία, συνεργάστηκαν άψογα μεταξύ τους. Ήταν ε, η συνεργασία σε εθελοντική βάση και μέχρι σήμερα πάντα κατάφερναν να αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα παρουσιαστεί. Να σας δώσω και το παράδειγμα της Γαλλίας και τι γίνεται με τις όμορες χώρες. Το blackout στην Ιταλία που προκλήθηκε από το γεγονός που είναι μεγάλο εισαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας η Ιταλία οδήγησε σε κάποιες άλλες λύσεις, δηλαδή διπλές γραμμές που μπαίνουν στο σύστημα κτλ έτσι ώστε να υπάρχει πάντα μια γραμμή διαθέσιμη σε περίπτωση blackout, σε περίπτωση downtime, ότι υπάρχει κάποια δυνατότητα να παρακαμφθεί το πρόβλημα, γιατί οι δύο ακριβώ γραμμέ το επιτρέπουν. Αλλά αυτό δεν είναι ρύθμιση από την αγορά την ίδια, είναι μέσω συνεργασία που το πετύχαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάρινς που είναι και εισηγητής για το επόμενο, για τους επόμενους δύο φακέλους ζητάει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή και είναι όντω ενδιαφέρον γιατί στι δικέ σου τροπολογίε ε, ήταν πολλά ενδιαφέροντα. Ήθελα να κάνω και ένα σχόλιο για τη συζήτηση. Ε, αναφέρθηκε στη Γαλλία. Και μας είπε πως όντως είναι χαοτική η κατάσταση και υπάρχουν προβλήματα. Νομίζω έχει να κάνει με το αν βλέπει κανεί το ποτήρι μισογεμάτο ή μισοάδιο. Σε επίπεδο καταναλωτή δεν συνέβη τίποτα. Γιατί οι TSO τελικά του έλυσαν το πρόβλημα. Και αυτό αποδεικνύει ότι τελικά Θα συμφωνήσω με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όντω θα έπρεπε να έχουν ε, καλύτερο σχέδιο έκτακτη ανάγκη εν κρίσεων. Αλλά το σύστημα τελικά κράτησε. Παρόλο που είχαν τεράστιε ε, αναταραχέ. Οπότε ήταν μια περίπτωση που ό,τι μπορούσε να πάει στραβά πήγε, αλλά παρόλα αυτά τα κατάφερε. Και νομίζω ότι η συγητή πολύ σωστά τονίζει ε, το ρόλο της ΕΝΙΣΑ και λέει θα πρέπει να συμβουλεύεται τους TSO πριν αναλάβει δράση γιατί ό,τι κανόνες και να έχουν και να λέμε ότι όταν ο πυροσβέστης ανέβει τη σκάλα την, για να ε, καταπολεμήσει τη φωτιά πρέπει να κρατάει τη μάνικα με τα δύο χέρια ε, την ώρα που θα ανέβει ο πυροσβέστης θα αποφασίσει με πόσα χέρια θα την κρατάει οπότε Εντάξει, καλύτερο συντονισμό μεν, αλλά η TSO να είναι μονίμως ενήμερη. Γιατί αυτοί είναι οι πυροσβέστε μας. Και όχι μόνο σβήνουν φωτιέ, αλλά το διαχειρίζεται το σύστημα και σε καθημερινή βάση. Οπότε δεν θα πρέπει εμεί ε, να ε, παρακάμψουμε το σύστημα, αλλά να το βελτιώσουμε. Άρα λοιπόν ο εισηγητή ε, νομίζω τα γράφει καλά. Ε, Ευχαριστώ πολύ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κ. Πόρχατ από την Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, Γενικό Διευθυντής. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, καταρχάς να υπογραμμίσω αυτά που είπε ο κ. Τούρμες και εν μέρη διαφωνώ μαζί σα, κύριε Κάρενς. Κοιτάξτε, έχουμε δύο παραδείγματα. Η Γαλλία ήταν ασφαλής διότι υπήρχε προκαθορισμένο σχέδιο για αμοιβαία αρρωγή. Στα νοτιοανατολικά συνέβη ακριβώς το αντίθετο. Ο καθένας κινήθηκε εγωιστικά και η Ρουμανία και η Βουλγαρία. Αν χρειαζόμασταν στοιχεία ότι ο κανονισμός για την προτεμασία του κινδύνου θα έπρεπε να υπάρξει, τα στοιχεία μας τα έδωσε ο Ιανουάριος. Σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζουμε την ε, έκθεση που υπευλήθη και τις τροπολογίες. Οι τροπολογίες σε πολύ σημαντικό βαθμό οδηγούν σε περαιτέρω διευκρινήσεις και σε ενίσχυση του κειμένου. Να αναφερθώ στην ε, εμπιστευτικότητα ευαισθήτων πληροφοριών. Χρειάζεται ενίσχυση το κείμενο εκεί. Συμφωνούμε με την τροπολογία ότι η εμπιστευτικότητα ευαισθητών πληροφοριών που σχετίζονται με κακοήθεις επιθέσεις ε, πρέπει να είναι κάτι που διαφυλάσσεται σε όλες τις φάσεις. Στηρίζουμε τη σχετική τροπολογία. Το ίδιο ισχύει ε, όσον αφορά το βελτιωμένο ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το συντονισμό όσον αφορά περιφερειακές συμφωνίες και σχετικά με τους μηχανισμούς συνεργασίας με τα χαράς να αναλάβουμε αυτό το ρόλο κανένα πρόβλημα επίσης με τις τροπολογίες σας που αφορούν τις προθεσμίες διότι μπορούμε να τις δεχτούμε όλες. Δεν θα οδηγήσουν σε παράταση και επέκταση τελικής ε, ημερομηνίας. Μια προειδοποίηση όσον αφορά την αμοιβαία αρρωγή. Εκεί προτείνεται διαφορετική διατύπωση. Λέτε ότι η αμοιβαία αρρωγή θα υπόκειται σε σχήμα αποζημίωσης που καθορίζεται εκ των προτέρων. Με αυτή τη διατύπωση διαβλέπουμε έναν κίνδυνο. Τι θα συμβεί αν το όλο αυτό σχήμα δεν προκαθοριστεί. Σημαίνει ότι η αμοιβαία αρρωγή δεν θα εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Γι' αυτό σας καλώ να επανεξετάσετε το κείμενο με τη δική μας διατύπωση αμοιβαία αρρωγή με την επιφύλαξη αποζημίωσης. έχουν πιο γενική προσέγγιση. Αν μπορείτε να το αποσαφηνίσετε το κείμενο. Δεν θέλετε, ε, αν δεν υπάρχει συμπεφωνημένο ε, σύστημα αποζημίωσης, να μην υπάρξει αμοιβαία αρρωγή. Χρειάζεται ευκίνηση το κείμενο. Τελικό σχόλιο για περιφερειακή συνεργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή. Όχι όσο αφορά την προετοιμασία του κινδύνου για το σχεδιασμό και της αγοράς, κάτι που θα συζητηθεί αργότερα. Έχουμε αυτές τις δύο λειτουργίες που προβλέψαμε στο σχεδιασμό της αγοράς και την πρόταση για την προετοιμασία και αντιμετώπιση κινδύνων. Έχουμε εντοπισμό ενδεχομένων κρίσεως και αιτήσια προσωμείωση κρίσεων. Πιστεύω ότι αν αφαιρέσουμε αυτές τις ε, λειτουργίες από το σχεδιασμό της αγοράς, ας γίνει έτσι. Αλλά για την προετοιμασία αντιμετωπίσεως κινδύνων θα πρέπει αυτές οι πτυχές να παραμείνουν, διότι οι αιτήσιες ε, προσωμιώσεις και ο εντοπισμός ενδεχομένων κινδύνων είναι πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία για να προετοιμαζόμαστε κατάλληλα για το χείριστο των, στην κρίσεων. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ κύριε Γενική Διευθυντά σαφής οι θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ πολύ. Ο εισηγητής μας, ο συνάδελφος Ανωνάτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Άκουσα παρεμβάσεις πολύ λογικές και μπορώ να συμφωνήσω μαζί τους. Μπορούμε να συνεργαστούμε συντονισμένα και γρήγορα και να οδηγηθούμε σε θετικότατο αποτέλεσμα και τελευταίες σκέψεις του εκπροσώπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θεώρησα ότι ήταν πάρα πολύ λογικές και θα ληφθούν υπόψη. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει ιδεολογική ακαμψία, οπότε μέσω συνεργασίας θα βρούμε λύση ε, η οποία θα τύχει μια ευρεία υποστηρίξεως. Αυτό πιστεύω και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. 37 δευτερόλεπτα. Υπέροχα. Όλοι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι πριν τις διακοπές, υπέροχα. Μετά τις διακοπές ελπίζω να είμαστε στην ίδια κατάσταση. Προθεσμία η αποβολή τροπολογιών. Καλά μαντάτα για όλους σας. 13 Σεπτεμβρίου. Όχι όπως πριν, αρχές Σεπτεμβρίου, τώρα μέσα Σεπτεμβρίου. Πολύ, πολύ καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ψηφοφορία στην Επιτροπή μας θα λάβει χώρα τον μήνα Δεκέμβριο. Στρεφόμαστε τώρα σε σημαντικό θέμα δύο ζητήματα. Εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και κοινή κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κανονισμός και οδηγία. Γενικώ πώς Έχουν πρόταση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή, μετάδοση, πώληση, αγορά και κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Αν θα πρέπει να είναι πιο πράσινη η ηλεκτρική ενέργεια, να βασίζεται στην αγορά, αν θα πρέπει να είναι αποδοτικότερη η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγή καταναλωτές, οι prosumers. Ε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η και για τα δύο θέματα είναι ο συνάδελφος Κάρινς Έχουμε τους ίδιους σκιώδες συγκητές και τα δύο αυτά θέματα έχουν πολλά αλληλένδετα ζητήματα. Ήταν καλύτερο και ασφαλέστερο να εξεταστούν ομού. Ο εισηγητής πρότεινε 187 τροπολογίες, 129 για τον κανονισμό και 58 για την οδηγία. Συνάδελφε, Καρίνς, Κριστιανής, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ. Εμένα μου άρεσε τόσο πολύ η πρόταση Κομισιόν που είπα να την ενισχύσω λίγο. Η... Το νομοθέτημα αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς εμείς οι νομοθέτες μπορούμε να επιτύχουμε χαμηλότερες τιμές τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τα νοικοκυριά και σε ένα πλαίσιο ε, παγκόσμιου ανταγωνισμού όσο χαμηλότερη είναι η τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο ανταγωνιστικότερες είναι βεβαίως και οι επιχειρήσεις. Η Κομισιόν λοιπόν υιοθετεί μια προσέγγιση που βασίζεται στην αγορά και αυτή την προσέγγιση θα ήθελα εγώ ε, με τις προτάσεις μου να ενισχύσω. Να μην υπάρχει όριο χονδρικής ε, αγοράς. Ε, είναι σημαντικό αυτό το στοιχείο, αν θέλουμε εύρυθμες αγορές. Για τις δυναμικότητες έχω, έχουμε πει ότι θα πρέπει να είναι έσχατο μέσο αφού εξαντληθεί η περιφερειακή συνεργασία και εφόσον διαπιστωθεί ότι οι φορείς της αγοράς δεν μπορούν να εξασφαλίσουν ε, την ε, επάρκεια της τροφοδοσίας. Αλλά στόχος πρέπει να είναι ε, παραγωγή εφεδρική η οποία θα αξιοποιείται όποτε χρειάζεται. Επίσης, πρέπει να εξισορροπηθούν οι ευθύνες όλων των, των εμπλεκόμενων φορέων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένας τρόπος για να εξασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της ε, αγοράς. Όταν κάποιος λοιπόν πουλά ηλεκτρική ενέργεια σε κάποιον άλλον και τελικά η ηλεκτρική ενέργεια αυτή δεν είναι διαθέσιμη, τότε θα πρέπει τα στρατηγικά αποθέματα να αξιοποιούνται. Ο καταναλωτής βεβαίως δεν διαπιστώνει ποτέ ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά ο πολιτής είτε είναι παραγωγός, είτε είναι εγκατάσταση αποθεματοποίησης ε, θα καταβάλει το τίμημα. Όποιο και αν είναι αυτό. Αυτός είναι ένας κανόνας απαραίτητος προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι ο πολιτής ηλεκτρικής ενέργειας θα πουλά μόνο αυτά που ξέρει ότι ε, θα έχει στη διάθεσή του μειώνοντας έτσι και την ανάγκη ε, στο μέλλον για την δημιουργία δυναμικότητας και αποθεματοποίησης. Διότι αν έχεις κάνει λάθος θα το λάβεις υπόψη σου την επόμενη φορά. Νομίζω ότι ε, αυτό ε, αντικατοπτρίζεται και στις τροπολογίες μου. Για τις ζώνες υποβολής προσφορών πρέπει ομόφωνα να λαμβάνεται η απόφαση από τα ε, κράτη-μέλη ε, όταν δεν μπορεί να ληφθεί η απόφαση, ωστόσο, θα πρέπει να παρεμβαίνει η Κομισιόν, η οποία και θα λαμβάνει την τελική ε, απόφαση για τη δημιουργία μιας ε, ζώνης υποβολής προσφορών, ώστε το κράτος μέλος και η Κομισιόν να έχουν την, την δυνατότητα να βρουν την σωστή λύση ε, για να αποφευχθεί ε, η συμφόρηση με την κατασκευή και νέων αγωγών. Τρίτον, ε, δεν συμφωνώ με την πρώτη της Κομισιόν για τα περιφερειακά, κέντρα, τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα. Έχω εδώ στις Βρυξέλλες συζητήσει αρκετές ώρες συζητώντας με TSO, με ρυθμιστικές αρχές και ε, είμαι απόλυτα πεπισμένος για την ανάγκη ενίσχυσης συνεργασία σε επιχειρησιακό ή άλλο επίπεδο. Ωστόσο, δεν πρέπει να μπλέκουμε ανώμια πράγματα. Η ευθύνη για τη λειτουργία των δικτύων ε, εναπόκειται στους TSO. Αυτό όμως δεν αποκλείει την καλύτερη συνεργασία. Λοιπόν, προτείνω ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, αλλά περιφερειακά συντονιστικά κέντρα. Όταν θα ε, κατακτήσουμε την ε, ομόσπονδη Ευρώπη, τότε μπορούμε να προχωρήσουμε και σε κάτι τέτοιο. Αν όμως αυτός ο στόχος δεν επιτευχθεί, τότε θα πρέπει να επιλέξουμε τη δεύτερη καλύτερη λύση. Δηλαδή, κυρίαρχα κράτη-μέλη τα οποία θα έχουν τα TSO τους και με τους οποίους αυτά τα κράτη-μέλη θα συνεργάζονται. Και αυτό είναι και μια ανάγκη που προκύπτει από την ίδια την καθημερινότητα και από την ίδια την ζωή. Αντί λοιπόν να υπάρχουν βρόχοι που θα διέρχονται μέσα από την ε, Γερμανία για παράδειγμα και θα πρέπει κάθε μέρα να αντιμετωπίζονται κρίσεις, ε, αυτό είναι κάτι το οποίο είναι, είναι ε, ανάγκη βάσει των νόμων της, ε, της φυσικής. Γιατί οι νόμοι της φυσικής δεν συνάδουν πάντοτε με το που πηγαίνουν οι πωλήσει, ούτε ταυτίζονται αυτά τα δύο. Άρα, για μένα, ο συντονισμός είναι ε, σημαντικότερος και η ευθύνη να, εναπόκειται, να εξακολουθήσει να εναπόκειται στους TSO, δηλαδή τους ανθρώπους που θα πρέπει να εξασφαλίζουν τις ε, ροές της ηλεκτρικής ανέργειας. Να πω και κάποια λόγια για την οδηγία. Εδώ είναι σημαντικό η, ότι η αποθήκευση επίσης θα πρέπει να ρυθμίζεται από την αγορά. TSO και DSO δεν θα πρέπει να παρεμβαίνουν στο παιχνίδι εκτός αν δεν υπάρχει άλλη λύση. Θέλουμε δηλαδή ε, και η αποθήκευση να ε, αποτελέσει ε, κλάδο που θα ρυθμίζεται από την αγορά. Έχω υποβάλει κάποιες τροπολογίες και για τις ε, ζωτική σημασία πληροφορίε. Ναι, οι καταναλωτέ θα πρέπει να ενημερώνονται, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει κάθε εταιρεία να αποστέλει δεκασέλιδου λογαριασμού με περίτες πληροφορίε. Μπορεί σε ένα λογαριασμό να βάλει τι βασικέ πληροφορίε, τι, είναι, ε, τι πληρώνει για, την, για την ηλεκτρική ενέργεια, τι είναι φόρο, τι είναι ε, οι άλλες χρεώσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει λόγος να πλημμυρίζουμε και να υπερφορτώνουμε τους καταναλωτές με υπερβολικές προφορίες. Αυτά από μένα προσβλέπω στη συνεργασία με όλους τους κοιόδης στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις σας και για τις τροπολογίες σας, την έκθεσή σας. Η κυρία Βέρνερ, εκ μέρους των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Κάρινς για την εξαιρετική έκθεσή σας. Συμμερίζομαι την προσέγγισή σας σε πολλά σημεία, ιδίως όσον αφορά τους μηχανισμούς δυναμικότητας, τους ROCs και τα bidding zones και εδώ ε, μπορείτε να βασιστείτε στην υποστήριξή μου. Βεβαίως με κάποια άλλα θέματα διαφωνώ. Πρώτον, διαγράψατε την, ε, την προτεραιότητα ε, της διασύνδεσης και κάπως έχετε ε, και έχω μια διαφορετική ε, άποψη όσον αφορά τις ισορροπίες των ευθυνών. Θα υποβάλω όμως και σχετικές τροπολογίες. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι οι προτάσεις σας για τους μηχανισμούς δυναμικότητας είναι πολύ καλές, ιδίως όσον αφορά την ε, διασύνδεση μεταξύ των αποθεμάτων που πάνε στην αγορά και των στρατηγικών αποθεμάτων και νομίζω ότι είναι πολύ καλό το γεγονός ότι ο, στην τροπολογία 57 επισημαίνεται ότι θα πρέπει να ε, εξετάζονται άλλα κοστοποδοτικότερα μέτρη προτού αξιοποιηθούν ε, τα στρατηγικά αποθέματα. Βεβαίως το ζήτημα αυτό έχει ε, σχέση και με την ενεργειακή μετάβαση. Φυσικά η ηλεκτρική ενέργεια και η αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να απαλλαγεί από τον άνθρακα, αλλά θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι εργαζόμενοι, οι περιφέρειες, που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τον ε, λιγνίτη και από τον άνθρακα. Πρέπει λοιπόν η διαδικασία αυτή να προσαρμοστεί και σε αυτή την πραγματικότητα. Πολύ καλό θεωρώ επίσης το γεγονός ότι αναφέρεστε στα WOPs και το γεγονός ότι τα μετονομάζεται σε ε, περιφερειακά ε, κέντρα συνεργασίας γιατί δεν έχουν σχέση με το επιχειρησιακό κομμάτι άμεσα αυτά τα κέντρα και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και επίσης βρίσκω σημαντικό το γεγονός ότι αναβαθμίζεται αυτά τα κέντρα σε συντονιστικά ώστε να μην δημιουργούνται παράλληλες δομές αλλά ώστε να βασιστούμε σε αυτά που ήδη υπάρχουν. Επίσης είναι σημαντικό οι διατάξεις αυτές να ψηφιστούν κατά την ε, συνήθεια νομοθετική διαδικασία και όχι μόνο μέσω των κωδικών δικτύων. Ε, δική μου θέση είναι επίσης ότι ε, είναι πολύ σημαντικό οι WOCs να αποκτήσουν και αρμοδιότητα λήψη αποθάσεων. Επίσης, συμφωνώ με τον άποψη του κυρίου Κάρνς για τη διεύρυνση των ζωνών θεωρώ ότι οι μικρές ζώνες δεν ε, ε, ε, αποφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα όπως, φαίνεται, φάνηκε και στην Σουηδία. Επίσης συμφωνώ ότι και οι μικροί DSO θα πρέπει να εκπροσωπούνται. Κάποια ερωτηματικά έχω όσον αφορά την, την, το θέμα της αξίας των χαμένων φορτίων, δηλαδή μια θεωρητική υψηλή τιμή που είναι διατεθειμένοι οι να, να καταβάλουν, κάτι όμως που μπορεί να οδηγήσει σε απολεσθέντα φορτία. Κάτι τέτοιο μπορεί και να οδηγήσει σε στρέβλωση της αγοράς, αλλά δεν έχω καταλήξει ακόμα οριστικά. Επίσης, κάτι που είναι σημαντικό για μένα και την ομάδα μου. Ε, πρέπει να εξασφαλιστεί ε, η, η προτεραιότητα για την εισαγωγή και τη διασύνδεση ε, ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Θεωρείτε όμως, κύριε Κάρενς, ότι η αγορά ήδη λειτουργεί εύρυθμα και ότι ε, όλοι οι φορείς και οι εμπλεκόμενοι έχουν δίκαιη πρόσβαση στην αγορά και στα δίκτυα. Κάτι τέτοιο όμως, κατά τη γνώμη μου, δεν ισχύει. Γι' αυτό και εμείς ως ομάδα επιμένουμε στην υποστήριξη και την ενίσχυση των ΑΠΕ. Όπως άλλωστε υποστηρίζονται και ενισχύονται και ο άνθρακας και η πυρηνική ενέργεια. Επίσης, στην παράγραφο 4 συμφωνώ μαζί σας ε, ε, σε πολλά θέματα. Ωστόσο, όσον αφορά την ενεργειακή ένδια, την προστασία των καταναλωτών και τις ενεργειακές κανότητες, νομίζω ότι είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε σε μεγαλύτερο βάρος Συμφωνώ με αυτό που είπατε για τις 24 ώρες, να υπάρχει αυτό το χρονικό περιθώριο. Ωστόσο, όσον αφορά τα ε, συγκριτικά εργαλεία, πιστεύω ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να καθιστούν τα συστήματά τους ακόμη πιο φιλόδοξα. Συμφωνώ λοιπόν μαζί σας εδώ ότι θα πρέπει να υπάρχουν ελάχιστες απαιτήσει, όμως υπάρχουν και κάποιες ε, προσεγγίσεις δικές σας με τις οποίες διαφωνούμε. Εσείς στην ενεργειακή ένδια, για παράδειγμα, θεωρείτε ότι πρωτεύοντα λόγο θα πρέπει να έχουν τα εθνικά κοινωνικά συστήματα. Εμείς πάλι πιστεύουμε ότι θα πρέπει να προβλέπονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο διατάξεις που θα προστατεύουν αυτά τα, νοικο, νοικοκυριά. Ρυθμισμένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, αυτές βεβαίως ε, δεν ε, συνάδουν με την, ε, με, με την θέση στο επίκεντρο της αγοράς. Ωστόσο, ε, νομίζω ότι και εδώ θα πρέπει να ε, εισαχθούν ορισμένα κοινωνικά κριτήρια, διότι δεν είναι δυνατόν ο διευθυντή μια τράπεζα, για παράδειγμα, να πληρώνει την ίδια τιμή με, με, με την κομμότρια που πληρώνει ε, τον λογαριασμό της ηλεκτρικής ενέργειάς της. Ο πρόεδρο διακόπτει την ομιλήτρια και τη επισημαίνει ότι έχει υπερβεί τον χρόνο που είχε στη διάθεσή της. Σας, ζητώ συγγνώμη και ολοκληρώνει η ομιλήτρια. Επίσης, για τη διαμεσολάβηση και την επίλυση διαφορών, συμφωνώ με, αυτό που λέτε, πρέπει να διατηρηθεί το σύστημα που προβλεπόταν στην, στην προηγούμενη ε, ε, οδηγία για τις, για, για τις μορφές των δεδομένων Νομίζω και εγώ ότι πρέπει πρώτα να εξασφαλιστεί, να, ε, καθοριστεί αυτό το θέμα σε εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια να υπάρξει μια εναρμόνιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Okay. Um, next speaker. Επόμενος ομιλητής, ο κ. Χρυστοδέμσκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να συνταχθώ με όσους έχουν ευχαριστήσει τον κύριο Κάριντς. Πιστεύω πως η συνεισφορά του είναι εξαιρετικά χρήσιμη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ συνεκτική η προσέγγιση που ακολουθεί και σε πάρα πολλά σημεία νομίζω πως μιλάμε την ίδια γλώσσα. Για παράδειγμα, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού, και άλλα σχετικά. Υπάρχει βέβαια ένα σημείο στο οποίο δεν έχω την ίδια άποψη ε, με τον κύριο Κάριντς. Και το σημείο αυτό είναι το κατά πόσο μπορούμε να χρησιμοποιούμε και να καταφεύγουμε στην αγορά για να μας λύσει όλα τα προβλήματα σε έναν κλάδο ο οποίος βασίζεται πάρα πολύ σε ενισχύσεις και επιδοτήσεις και όπου η αγορά έχει ένα μάλλον περιορισμένο ρόλο στα όσα γίνονται. Θέλω να σας δώσω κάποια παραδείγματα. Για παράδειγμα, η ηλεκτρική ενέργεια η οποία παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί εκεί πως χρειάζεται ρύθμιση. Αλλά νομίζω ότι πρόκειται για ένα πολιτικό σχέδιο, είναι ένα, μια πολιτική ιδεολογία που μας οδηγεί στη χρήση των ανανεώσιμων και στην καθαρή ενέργεια και αυτό είναι ένα στοιχείο που πρέπει να λάβουμε υπόψη. Υπάρχουν και άλλα θέματα με τα οποία θα δυσκολευτώ να συμφωνήσω και θα σας πω πως ο μηχανισμός δυναμικότητας για παράδειγμα είναι ένα θέμα με το οποίο εμείς αντιμετωπίζουμε πρόβλημα, όπως επίσης και οι αγορές ενέργειας, η τιμολόγηση ε, που γίνεται χοντρική η κατανομή αρμοδιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το πώς αυτή απηχείται ε, με το σχεδιασμό αυτών των ε, περιοχών τιμολόγησης, με τις ζώνες τιμολόγησης δηλαδή έχουμε πρόβλημα και πιστεύω πως θα βρούμε κάποιους συμβιβασμούς έτσι ώστε να μπορέσουμε κι εμείς με αποτελεσματικό τρόπο να διαπραγματευτούμε και με το Συμβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κάλλας. Η κυρία Κάλλα, με συγχωρείτε, ευχαριστώ πολύ ε, τον εισηγητή για τι δύο αυτέ εκθέσει και πρέπει να σα πω πω αυτή η φάκελη είναι μεγάλη. Έχουμε συζητήσει ήδη το χρονοδιάγραμμα, οπότε υπάρχουν μόνο κανένα δύο θέματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Καταρχήν, χαιρετίζω στα τα σχέδια έκθεση, γιατί σε μεγάλο βαθμό ενισχύουν την προσέγγιση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που βασίζεται στην αγορά και θεωρώ πως αυτό είναι σημαντικό γιατί η στρέβλωση της αγοράς οδηγεί σε μη αποδοτικές αγορές και αυτό επηρεάζει τους καταναλωτές γιατί τελικά επιβάλλει ψηλότερο κόστος στην ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης στηρίζω τον εισηγητή γιατί λέει πως δεν πρέπει πια να έχουμε διατίμηση στις τιμές, ε, θα πρέπει να ξεχωρίσουμε την ενεργειακή πολιτική από την κοινωνική πολιτική και καλωσορίζω τα όσα ο, λέει ο εισηγητής για να μπορούν να αλλάξουν πάροχο εύκολα και να σας πω πως είναι οι πιο ευάλωτες ομάδες που τελικά δεν μπορούν να απαλλαγούν από τα πιο ακριβά συμβόλαια. Αλλά είπαμε, θα μπορεί να αλλάξει κανείς από το 2025. Όχι, γιατί να περιμένουμε, ας το κάνουμε και νωρίτερα. Επίσης, χαιρετίζω την προσέγγιση του εισηγητή για το μηχανισμό δυναμικότητας, γιατί νομίζω ότι τα σημεία τα επόμενα θα πρέπει να είναι ξεκάθαρα, να είναι στην νομοθεσία, να μιλήσουμε για το διαχωρισμό και για όλα τα παρακάτω. Και γιατί ο εισηγητής μιλάει για το όριο των 450 μόνο πέντε χρόνια μετά ε, την θέση σε ισχύ της νομοθεσίας τώρα για τους aggregators εγώ δεν κατάλαβα ακριβώς χαιρετίζω την προσπάθεια αλλά δεν κατάλαβα καλά τι γίνεται με την αποζημίωση δηλαδή το κείμενο δεν είναι σαφές. Καταλαβαίνω πως οι aggregators θα πρέπει να κάνουν μια ε, ισορροπημένη ε, προσπάθεια να ικανοποιήσουν τη ζήτηση. Αλλά αν κατάλαβα καλά, αυτό είναι οι aggregators που πολλούν την ζήτηση την προηγούμενη μέρα ή κάνουν συμφωνίες την προηγούμενη μέρα και πολλούν την ε, ζήτηση την επόμενη μέρα. Δεν έχω καταλάβει ακριβώ πώ γίνεται και γι' αυτό δεν καταλαβαίνω ακριβώ Πού μπαίνει το κομμάτι της αντισταθμητικής ε, αποζημίωσης. Αυτό θα δούμε να με εξηγήσετε. Επίσης, περιφερειακή συνεργασία. Δεν πιστεύω πως η ενισχυμένη περιφερειακή ε, συνεργασία θα λάβει η χώρα αν ε, τα κέντρα δεν έχουν, τα περιφερειακά κέντρα συντονισμού δεν έχουν τη δυνατότητα λήψης απόφασης. Ξέρουμε που είναι τα σημεία συμφόρησης. Είναι εκεί όπου δεν υπάρχει καλή συνεργασία. Εκεί που υπάρχει δεν χρειάζεται έχουμε πρόβλημα με τα σημεία στα οποία η συνεργασία δεν λειτουργεί και έχουμε και ένα θέμα με τους περιφερειακούς παίκτες γιατί πιστεύουμε ότι και αυτοί θα πρέπει να ε, έχουν το λόγο τους. Αυτές οι συστάσεις τι νόημα έχουν αν θέλουμε να εμβαθύνουμε στην ενιαία αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Τούρμες, εκπροσωπώντας τους πρασίνους, βλέπω την έκθεση αυτή ας μια έκθεση η οποία σε τεχνικό επίπεδο έχει γραφτεί σωστά, σας συγχαίρω. Έχει μια φιλελεύθερη προσέγγιση, αλλά ίσως λίγο λέω φιλελεύθερη κατά καιρού. Καλή πρόταση για το μηχανισμό δυναμικότητας, για το απόθεμα σταθερότητας που θα είναι ένα πιο φθηνό σύστημα, 550, σωστό νούμερο, αλλά γιατί αποδυναμώνει την ευρωπαϊκή διάσταση με την περιφερειακή ζώνη και με, τους με, τις... Ε, με την περιφερειακή συνεργασία και τις ζώνες δημοπράτησης. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί να μην ενισχύσουμε τους aggregators, για παράδειγμα, μια και αποτελούν προϋπόθεση, έτσι ώστε οι αλγόριθμοι αυτοί ε, να ενεργοποιούν ε, τους καταναλωτές και τους πολιτές και γιατί να αποδυναμώσουμε τις ενεργειακές κοινότητες και γιατί να μην ε, τονίσουμε την ανάγκη για επένδυση ε, στις ΑΠΕ. Δηλαδή ε, αναδρομικές αλλαγές, αναδρομικές αλλαγές. Εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, να αποδυναμώσουμε επενδύσεις οι οποίες έχουν ήδη γίνει. Εμείς αυτό το καταγγέλουμε συνήθως. Και μετά υπάρχει το θέμα της ισόρροπης ευθύνης. Αν όλες οι αγορές ήταν τόσο ρευστέ, όπω η αγορά και είχαν τόσους παίκτε, τότε ναι, θα μπορούσαν να έχουν πολύ μεγαλύτερη ε, υποχρέωση που η για τι ΑΠΕ. Αλλά ακόμα και στη Γερμανία πολύ μικροί παίκτε προστατεύονται. Γιατί? Γιατί οι γερμανικές αρχές μετά από πάρα πολλά χρόνια ε, ανάπτυξης πιστεύουν πως η αγορά ακόμα δεν έχει οριμάσει έτσι ώστε να μπορεί κάθε μεμονωμένο παίκτη να αναλάβει τι ευθύνε του. Και όπω λέει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, του μικρού παίκτε πρέπει να του προστατεύσουμε. Και νομίζω πω για την προτεραιότητα στην πρόσβαση για τις ΑΠΕ στην Ευρώπη τα νοικοκυριά ακόμα δεν είναι έτοιμα. Δεν μπορούμε να έχουμε μια έτσι ξεκάθαρη λύση κατά αποκοπή. Όχι, την αντίστροφη λογική πρέπει να ακολουθήσουμε. Μια σειρά από όρους για το πότε και όταν η αγορά θα είναι έτοιμη και όχι με έναν άδικο τρόπο. Γιατί το αποτέλεσμα τελικά θα είναι περισσότερο ρίσκο, περισσότερο κόστος επενδυτικό, περισσότερο κόστος στον καταναλωτή. Δηλαδή, 90% συν στις ανανεώσιμες. Θα το υποσκάψουμε αυτό. Μα τότε μόνο το κόστος θα αυξήσουμε. Και για τα υπόλοιπα να σας πω ότι υπάρχει ένα θέμα στο οποίο δεν έχετε κάνει τη δουλειά σας και αυτό είναι η δίκαιη αγορά. Πού είναι το άνοιγμα στην αγορά και η έκθεση στην αγορά της πυρηνικής ενέργειας. Κάνετε κάτι σε αυτό. Δεν πληρώνουν ασφάλεια, δεν ε, ε, έχουν καθόλου ε, αποθεματικό για την αποξύλωση. Τι συμβαίνει εκεί. Τώρα και για τη διαφορά μεταξύ χονδρική και λιανιβουρίου. και να προστατεύσουμε του μικροκτανολίτες. Χθε το πρώτο πάνελ, η πρώτη συνεδρία ήταν πολύ ενδιαφέρον. Και τι μα είπε ο άνθρωπο από την Εστονία. Θέλουμε μαζικά να έχουμε ευφυείς μετρητές, αλλά αυτό που έκανε τους εστονούς να πληρώνουν λιγότερο είναι η οροφή. Η οροφή από την οποία και πάνω μπορεί ή όχι ένας λιανέμπορος ηλεκτρικής ενέργειας να πουλήσει ηλεκτρική ενέργεια. Νομίζω λοιπόν ότι όταν συζητάμε τα θέματα αυτά πρέπει να δούμε. Θέλουμε τις ρυθμιζόμενες τιμές να τις καταργήσουμε. Όχι! Θέλουμε να μην επιτρέπουμε την κερδοσκοπία. Και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι αυτοί που δρούν στο λιανικό εμπόριο θα κερδίσουν κάτι από τους καταναλωτές που είναι όχι πολύ καλά καταρτισμένοι, όχι, είναι λίγο τεμπέληδες. Και τέλος, το μελλοντικό σύστημα θα είναι πάρα πολύ αποκεντρωμένο και οι περισσότερες από αυτές τις συνδέσεις θα γίνονται σε DSO επίπεδο. Άρα οι DSO θα γίνουν όλο και πιο σημαντικοί ως ουδέτερη πλατφόρμα. Οπότε και αυτά θα πρέπει να τα συζητήσουμε, μια και ο, ο εκτελεστικός διευθυντής του δικτύου της Εστονίας μίλησε για την ουδετερότητα, γιατί δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε καινούργια ολιγοπόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ηλικιώτης παρακαλώ, εκ μέρου τη κυρία Έρνστ από την ΚΟΕ. Η Σκιώδη δεν μπορούσε να έρθει σήμερα και γι' αυτό μου ζήτησε να την αντικαταστήσω για την εσωτερική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί όλα αυτά έχουν ως σκοπό να εξασφαλίσουν μια ασφαλή μετάβαση του η πρόοδος θα καθυστερήσει και θα γίνει πιο δαπανηρή για τα κρατη με αυτά που προτείνεται και για τους λόγους αυτούς. Πιστεύουμε πως η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Περιφερειακά Συντονιστικά Κέντρα είναι καλή. Και οι αναφορές που γίνονται σε αυτά θα πρέπει να διατηρηθούν Χαιρετίζουμε το σχέδιο έκθεσης στο σημείο που αναφέρει πως ο μηχανισμός δυναμικότητας θα πρέπει να εισαχθεί ως μόνο μέσω ίστατης ανάγκης και καλό θα, πρέπει, θα ήταν να κράτη-μέλη να μας εξηγήσουν πώς χρησιμοποιούν άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα η αποθεματοποίηση, η απόκριση σε επίπεδο ζήτησης και η ενεργειακή αποδοτικότητα για να ελαφρύνουν όλα τα προβλήματα που έχουμε απαντήσει. Επίσης χαιρετίζουμε τον εισηγητή που διατηρεί αυτά τα κριτήρια επιλεξιμότητας για τη συμμετοχή στο, στο μηχανισμό δυναμικότητας με τα 550 ε, ε, γραμμάρια εκπομπών άνθρακα ανά κιλοβατόρα και νομίζω πως είναι απόλυτο απαραίτητο αυτό να ε, εφαρμοστεί για, όλες τις, για όλους τους σταθμούς παραγωγής μόλις τεθεί σε ισχύ νομοθεσία. Και τέλος θα πρέπει να δούμε και το θέμα το τι γίνεται με το δυναμικό βρώμικης ενέργειας που υπάρχει από θυματοποιηθεί. αυτό δεν, δεν αναφέρεται καθόλου. Και να σας πω πως έχουμε το σύστημα ανταλλαγή εκπομπών που δεν έχει δώσει τα μηνύματα ε, που θα μας επιτρέψουν να αποχωρήσουμε από την άνθρακα, οπότε θα πρέπει το θέμα αυτό της βρώμικης ενέργειας να το δούμε, γιατί το phasing out θα πρέπει να το διαχειριστούμε σωστά και έτσι ώστε να έχουμε μια δίκαιη μετάβαση για τις κοινότητες και τους εργαζόμενους που θα επηρεαστούν για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη σχετική οδηγία, ως σκιώδης μας θεωρεί πως χρειαζόμαστε οι νέες πηγές ενέργειας να θεωρηθούν προτεραιότητα στην πρόσβαση Και αυτό το priority dispatch για τις νέες ΑΠΕ θα πρέπει όντως να διατηρηθεί, αλλά τα όσα λέει η Κομισιόν δεν μπορούν να μας βρουν σύμφωνα όταν μιλάμε κυρίως για α, αναδρομικές αλλαγές, γιατί εδώ αυξάνει το κόστος της μεταβατικής περίοδου και θα πρέπει οι επένδυτες να θεωρήσουν πως είμαστε ένα σταθερό επενδυτικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ. Χρειαζόμαστε περισσότερες διευκρινήσεις για τις κοινότητες ενέργειας, οι οποίες κατά τη γνώμη μας αυτή τη στιγμή δεν αναγράφονται επαρκώς στην έκθεση. Θα πρέπει να δούμε τι σημαίνει τοπικές ενεργειακές κοινότητες, ποιος είναι ο ορισμός, να δούμε πώς μπορούν αυτές να μπουν στο σύστημα των λειτουργικών κοινοτήτων και δικτύων και θα πρέπει να έχουμε ίσως κανόνες για όλους, να το επιβάλλουν αυτό οι ρυθμιστές με διαφάνεια για τον καταναλωτή, για τις πράσινες προσφορές των ε, προμηθευτών. Ευχαριστώ. Thank you very much, Ευχαριστώ πολύ, συνάδελφα. Και ο κ. Ταμπουράνο, εκ μέρους του EFDD, σκιώδης εισηγητής, αλλά και συντονιστής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνούμε με την πρόθεση του εισηγητού να δημιουργήσουμε πραγματικά μια ισότιμη αγορά που θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους για τη να έχουμε χαμηλότερε τιμέ και ανταγωνιστικέ τιμέ του καταναλωτή, εγγυόμενοι ταυτόχρονα τον ασφαλή εφοδιασμό. Να υπενθυμίσω ότι πρέπει τα ανθρώπινα όντα να είναι στην πρώτη θέση και όχι η αγορά. Η αγορά είναι μόνο ένα εργαλείο για να πετύχουμε τον απότερο στόχο της ισότιμης διανομής των κοινωνικών αγαθών, όπως είναι το περιβάλλον, η υγεία, το κλίμα δεν θα πρέπει να δώσουμε στην αγορά ε, να τη θεωρήσουμε σαν μια νέα θεότητα και να ρυθμίζονται τα πάντα την αγορά όπως την ηλεκτρική αγορά. Πρέπει να δημιουργηθεί πραγματική ισότιμη διανομή του αγαθού. Να αναγνωρίζουμε όμως και διαφορές και δυνατότητες που έχουν οι διάφοροι φορείς για να ε, πετύχουμε τους στόχους. Δεν θα πρέπει να ισχύουν όλοι οι κανόνες οι ίδιοι για όλους, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδιαιτερότητες. Υπάρχουν διάφορα στρατηγήματα που προτείνονται από τους μεγάλους φορείς για να φέρουν σε μια ανοιχτική θέση τους μικρότερους εμπορευόμενους και προσπαθούν να καθυστερήσουν τη μετάβαση προς μια παραγωγή αποκεντρωμένη με ανανεώσιμες πηγές ε, ενέργειας και μικρότεροι φορείς και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ε, θα πρέπει να ε, τελικά να δίνουν μεγαλύτερα κέρδη στην επικράτηση στην οποία δρεύουν. Μέχρι τώρα ε, οι επιδοτήσεις είχαν στηρίξει την πυρηνική ενέργεια και τα ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει να έχουμε νέα βέση για την αγορά. Να έχουμε σύστημα αποζημιώσεως και αντιστάθμισης και όλοι οι εμπορευόμενοι να είναι στις ίδιες συνθήκες. Όχι όπως τον προηγούμενο αιώνα που δεν είχαμε υπολογισμό ε, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών πριν. Πρέπει να λάβουμε υπόψη διάφορους παράγοντες και τα διάφορα προβλήματα αντιμετωπιστούν. Να μην είναι, να μην είναι σε μειονεκτική θέση ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρακαλούμε να μιλάτε πιο αργά, λέει ο Πρόεδρος, να διευκολύνετε τους διερμηνείς. Πηγαίνετε πιο αργά για να μπορεί να γίνεται σωστά η διερμηνία, παρακαλώ, ο Πρόεδρος. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι σε διαρθρωτική θέση και ανταγωνιστική μειονεκτική εδώ και δεκαετίες, λόγω των κανόνων. Αλλά είναι η τεχνολογία όμως η εναλλακτική, πολύ σημαντική να πετύχουμε τους στόχους τους γεωπολιτικούς και τους κλιματολογικούς έχει παραμείνει η προτεραιότητα ε, της προσπάθειας εισόδου να μπορούμε να βοηθήσουμε οι εταιρείε ανανεωσίμων να μπορούν στην αγορά. Για να μην αυξηθεί η εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου από την παραγωγή ενέργειας. Πρέπει να είναι λειτουργικοί οι ικανότητα που θεσπίζουμε. Ο εισηγητής επιδεινώνει την πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπής ζητώντας την εξάλληψη την αναδρομική των προτεραιοτήτων. Πώς θα έχουμε βεβαιότητα επενδύσεων? Ίσως δεν είναι όλες οι επενδύσεις ίσες. Είναι πιο σημαντικές οι επενδύσεις στον πυρηνικό τομέα και στον τομέα ορυκτών καυσίμων. Πρέπει να βοηθήσουμε τις μικρές επιχειρήσεις να μπορούν να έχουν πρόσβαση στην αγορά. Πρέπει να μειωθεί το διοικητικό άχθος κυρίως έναντι των οικογενειών, έναντι φορέων μικρομεσαίων. Η προτινόμενη ακύρωση θα θέσει εμπόδια για τους μικρούς παραγωγούς ε, με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ιδιαιτερότητες όσον αφορά την παραγωγή ενέργειας. Η προτινόμενη αλλαγή διαιωνίζει τα προβλήματα και τις διακρίσεις και δυσκολεύει την ε, είσοδο στην αγορά των μικρών φορέων. Δεν συμφωνούμε με το σύστημα αποζημιώσεων όσον αφορά τους aggregators. Δεν θα πρέπει να στην ζωή το παρελθόν και να το προστατεύουμε το μέλλον. Πρέπει να προσβλέπουμε προς το μέλλον απαλλαγμένοι από τα φαντάσματα του παρελθόντος. Αυτά και ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφε. Η κυρία Νίβλερ έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφο Κάρινς για την εξαιρετική πρότασή του. Συμφωνώ με πολλά από αυτά που περιλαμβάνονται στο σχέδιο έκθεσης του. Υπάρχουν όμως και ορισμένοι τομείς ε, που θα πρέπει να τους συζητήσουμε. Θέλω να αναφερθώ σε τρία θέματα. Πρώτον, μηχανισμοί δυναμικότητας. Ιδίως άρθρο 23 παράγραφος 4. Εγώ θα ήθελα να διαγραφεί η συγκεκριμένη παράγραφος. Δεν μου αρέσει αυτό το μπέρδεμα μεταξύ των μηχανισμών ε, δυναμικότητας και των στόχων ε, για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής. Δεν συμφωνώ με αυτό το 50, ε, τον αριθμό που υπάρχει εκεί. Βλέπω όμως ότι τελικά ο εισηγητής, ε, αν και είχαμε συμφωνήσει επ' αυτού, το επανέφερε στο σχέδιο έκθεση του. Ε, Παρ' όλα αυτά θα ήθελα να το ξανασυζητήσουμε. Ε, επίσης ε, έχω και ορισμένε αμφιβολίες για το κατά πόσο τελικά είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα τέτοιο μηχανισμό στην δυναμικότητα. Θα το ξαναδιαβάσουμε όμω και θα το ξανασυζητήσουμε. Δεύτερον, ε, περιφερειακά κέντρα συνεργασία δεν μου πολύ αρέσουν, πρέπει να σας πω. Θεωρώ ότι η πρόταση ε, του συγκητή να ε, συσταθούν συντονιστικά κέντρα είναι καλά. Ε, εγώ δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς αφορούσε αυτή η πρόταση των, για τα κέντρα συνεργασίας. Ούτε κατάλαβα τι θα προσέθετε κάτι τέτοιο. Η TSO έτσι και σε, σε περιφερειακό επίπεδο συνεργάζονται. μάλλον αντιστρατεύεται τους στόχους που έχουμε θέσει το να δημιουργηθούν τέτοια κέντρα συνεργασίας γιατί δυσκολεύουν τελικά την, ε, την ε, εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. Και για τα bidding zones ε, νομίζω ότι και εδώ ο κύριος ε, Κάρινς έχει υποβάλει καλές προτάσεις, ιδίως ως προς το σκέλος που αναφέρει ότι τα κράτη-μέλη που πλήττονται θα πρέπει εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος να εξευρίσκουν μια κοινά αποδεκτή λύση. Εγώ διαφωνώ με το να παρεμβαίνει αυθαίρετα και αυτεπάγγελτα η Κομισιόν σε αυτές τις περιπτώσεις. Συμφωνώ με τον, με τον εισηγητή σε αυτό το θέμα. ευχαριστώ. πάρα πολύ, ο κύριος Λεβαντόφσκι. Ευχαριστώ. Συμφωνώ με τον Κριστιανής και με κάποιους άλλους ομιλητές. Ευπρόσδεκτη η προσέγγιση της οικονομίας της αγοράς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σχόλιο επιδόσεις, προδιαγραφές και τις Το αναφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το επαναλαμβάνει ο συγητής. Στην τροπολογία 63 και 550 κιλοβατόρες και εκπομπή διοξιδίου άνθρακος. Εδώ εξαλείφουμε τις περισσότερες μονάδες παραγωγής στη χώρα μου δεν βοηθάει ούτε μεταβατική περίοδος. Περισσότερο θα, πλειοψηφία θα έχουμε μονάδες παραγωγής από φυσικό αέριο και θα αυξήσουμε έτσι την εξάρτηση από εισαγωγή φυσικού αερίου. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Πολωνία, ίσως και για άλλες χώρες. Αυτό ίσως οδηγεί υψηλή τιμολόγηση δυναμικότητας. Άρα θα μετακυλιστεί αυτό σε κόστος για τους καταναλωτές. Καταβάλει προσπάθηση η Πολωνία να πετύχει τους στόχους για τις κλιματολογικές αλλαγές μέσω καθαρού άνθρακα και σχετικής τεχνολογίας. Αυτό είναι ανέφικτο με αυτού του είδους τις προδιαγραφές και τα πρότυπα που έχουμε στο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε. Επόμενος. Μπλάνκο Λόπεθ. Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για τη δουλειά που έκανε γιατί είναι δύο από τα ρυθμιστικά πλαίσια από τα πιο φιλόδοξα που αντιμετωπίζουμε. Και έχω ένα σχόλιο για το μηχανισμό δυναμικότητας. Να σας πω πως χρειαζόμαστε δυναμικότητα για να στηρίξουμε ένα σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας που θα βασίζεται σε ΑΠΕ. Αλλά αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρόφαση για να στηρίξουμε πηγές ενέργειας που ρηπαίνουν. Πιστεύω πως θα ήταν σφάλμα να καταργήσουμε την προτεραιότητα στην πρόσβαση και στο dispatching των ΑΠΕ. Και πιστεύω πως η πρόταση της ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι καλή και θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι ιδιαίτερες ε, συνθήκες των μικρών εγκαταστάσεων ΑΠΕ, όπως επίσης και οι εγκαταστάσεις που είναι πειραματικές και δεν είναι ανταγωνιστικές στην αγορά. Και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε πως δεν θα δοθεί προτεραιότητα στην, ηλεκτρική, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ρηπογόνων πηγών και αυτό εις βάρος της παραγωγής από ΑΠΕ. Και θα πρέπει για το σκοπό αυτό να υπογραμμίσουμε την ανάγκη για διασύνδεση έτσι ώστε να ε, εξελιχθεί μια πλήρως ολοκληρωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Και νομίζω η Ισπανία είναι ένα καλό παράδειγμα απομόνωσης. Η οδηγία αυτή αναφέρεται στην ανάγκη προστασίας των πολιτών που είναι ευάλωτοι. Θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καλύτερα τα μέτρα που θα πρέπει να λαμβάνονται για να αντιμετωπίζουμε το θέμα της ε, ανεργιακής Ευχαριστώ Ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ και εγώ τον συνάδελφο Κάρινς για την πρότασή του. Νομίζω ότι και μένα με ικανοποιεί πάρα πολύ. Αλλά τούτου λεχθέντος και συμμερίζοντας σε κάποιο βαθμό με τα όσα είπε ο συνάδελφος Μπλάνκο, για να γίνουν όλα αυτά, χρειάζεται να εφαρμόσουμε, ε, να χρησιμοποιήσουμε και κάποια εργαλεία που θα μας επιτρέψουν να εξελιχθούμε όχι μόνο στην Ιβερνική Χερσόνησο και σε άλλες χώρες. Υπάρχει πρόβλημα διασύνδεσης για να εξασφαλίσουμε πως θα έχουμε μια ροή ενέργειας η οποία θα είναι εγγυημένη και που θα εξασφαλίζει πως οι τιμές δεν έχουν μεγάλες διακυμάνσεις. Και επειδή θέλουμε να καταργήσουμε τις ρυθμιζόμενες τιμές, να δούμε πώς θα το καταφέρουμε αν δεν έχουμε τις απαραίτητες διασυνδέσεις. Το ίδιο θα λέγαμε και για το μηχανισμό δυναμικότητας, δηλαδή η αξιολόγηση για, τις, ε, για το δυναμικό θα πρέπει να λάβει υπόψη τι γίνεται με τις χώρες που είναι λίγο διασυνδεδεμένες. Θα πρέπει να επιμείνουμε και εκεί που θα πρέπει να βρούμε λύσεις είναι αυτός ο τύπος που θα μας επιτρέψει πραγματικά να δώσουμε κίνητρα για τις ΑΠΕ. Γιατί έχουμε χώρες οι οποίες χρειάζεται να διασυνδεθούν και που έχουν διαφορετικές πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούν και δεν έχουν, για παράδειγμα, το ίδιο ενδιαφέρον για τις ΑΠΕ, τότε οδηγούν σε μία ε, κατάσταση παγωμένη, η οποία είτε επιβραδύνει τη διασύνδεση, είτε δεν τη δίνει προτεραιότητα. Γιατί έτσι και το 10% που έχουμε βάλει λίγο είναι. Οπότε τελικά όλα οδηγούν στο πακέτο αυτό που είναι η διακυβέρνηση και τα λοιπά, να χρειάζεται να βρεθούν λύσεις που θα δώσουν κίνητρα οικονομικά, αποτελεσματικά για την ανάπτυξη των διασυνδέσεων ε, στο επίπεδο που πραγματικά χρειάζονται. Ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Κόχλιτσεκ. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου, τον κύριο Κάρεντς. Ευχαριστώ που κατανοήσατε ότι πρέπει να υπάρξει συντονισμός. Τα ETSOs πρέπει να γίνουν κέντρα συντονισμού. Αν γίνουν κάτι διαφορετικό, θα αλλάξουμε αυτό που ήδη λειτουργεί, αυτό που ισχύει και αυτό ποτέ δεν είναι καλή ιδέα. Οι βέλτιστες πρακτικές μας δείχνουν ότι αν κάτι λειτουργεί και θέλουμε να το αλλάξουμε, τότε αυτό θα καταρρεύσει. Όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια, γιατί να έχουμε αγορά, πρέπει να είναι διαθέσιμη η ηλεκτρική ενέργεια σε όλους. Είναι μια πρακτική απόφαση αυτή όπως και εξάλληψη της ε, ενεργειακής ένδειας. Είναι πολιτική απόφαση, είτε είναι στη Βαλτική το πρόβλημα, στην Πολωνία σε άλλα μέρη της ε, Ευρώπης. Είναι πάντα πιο δαπανηρό το να κάνουμε κάτι διαφορετικό, όπως το να ε, εγκαταστήσουμε καλώδια. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς διάνοια για να κάνει τον υπολογισμό. Δεν χρειαζόμαστε προτεραιότητες όσον αφορά την μεταφορά της ενέργειας. Σε περίπτωση κρίσης πρέπει να δούμε ποια είναι η προτεραιότητα. Αν έχετε μία κρίση με το φυσικό αέριο, τι πρέπει να κάνετε. Είναι να δώσετε θέρμανση στον πληθυσμό σαν προτεραιότητα. Δευτερευούση σημασία είναι να φροντίσετε τα δημόσια κτίρια σε αυτή την περίπτωση. Τρίτη θέση, ε, έχουν όλα τα άλλα. Δεν υπάρχει λοιπόν ανακαθορισμός προτεραιοτήτων, είναι πάντα σαφείς οι προτεραιότητες. Τι θα κάνει η κυβέρνηση, γιατί είναι υπεύθυνη η, κυβέρνηση. Στην τσεχική δημοκρατία καταφέραμε να εξηγιάνουμε κάποιες μεγάλες εταιρείες. Εγώ είμαι υπεύθυνο για την Baltic Energy. Εγώ ήμουν υπεύθυνο για κάποια ε, χαλιβουργία. Ε, τώρα παρέχει ενέργεια παράγει ενέργεια και μεταφέρει ενέργεια. Αλλά αυτό δεν είναι ευθύνη τη κυβέρνησης. Πρέπει να κάνουμε σωστή διάκριση. Αποθεματικό, δυναμικότητα. Χρειαζόμαστε μεγάλη δυνατότητα αποθεματοποίησης για τη Γερμανία Φερρυπίν, διαφορετική για άλλου. Πάντα όμως πρέπει κανείς να είναι σε θέση να καλύψει τι περιπτώσει blackout, blackout από φωτοβολταϊκά ή από ανεμογεννήτριες. Δεν είναι αξιόπιστες πηγές. Αυτό συνέβη πολλές φορές στην Γερμανία. Αν δεν έχεις λιακάδα, ε, δεν έχεις ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, αν δεν φυσάει άνεμος, δεν παράγουν οι ανεμογεννήτριες. Ε, αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο να το καταλάβει κανείς. Δεν είναι τίποτα δύσκολο. Ο κύριος Μπόρχαρτ από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με μια γενική παρατέρηση και για τις δύο εκθέσεις. Συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Τούρμες που είπε ότι και οι δύο εκθέσεις από τεχνική σκοπιά είναι πολύ καλές. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πιστεύω ότι η συνολική προσέγγιση που υιοθετείται σε αυτές τις δύο εκθέσεις καταδεικνύει ότι και τα δύο κείμενα ε, θέτουν ως στόχο τη μεγαλύτερη προστασία των καταναλωτών και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας. Και εδώ βεβαίως συμφωνούμε απόλυτα με την προσέγγιση αυτή που αποτελεί και την καθοδηγητική αρχή της δικής μας πρότασης. Και τέλος, βλέπω ότι και στις εκθέσεις και στις τροπολογίες εισάγονται και κάποιες νέες ιδέες για την ανάπτυξη πιθανών λύσεων. Ε, είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά που αναφέρθηκαν για τα bidding zones και η σχετική τροπολογία. Γιατί και είναι καλή διότι ε, καταδεικνύει ότι η διαμόρφωση αυτών των ζωνών δεν είναι μόνο τεχνική φύση ζήτημα, αλλά έχει και μια πολιτική διάσταση. Και γι' αυτό θεωρώ ότι είναι πολύ θετικό να δίνεται ε, στα κράτη-μέλη η δυνατότητα να διαμορφώνουν τις ζώνες αυτές και ως έσχατο μέσο να υπάρχει δυνατότητα ε, παρέμβασης κομισιών. Επίσης, εμείς ε, υποστηρίζουμε την ανάπτυξη των μηχανισμών δυναμικότητας και ε, συμφωνώ με αυτό που είπε ο εισηγητής ότι προσπαθεί να ενισχύσει την πρόταση της κομισιών. Πράγματι και εγώ την ίδια εικόνα έχω, την ίδια άποψη έχω σχηματίσει. Βεβαίως Υπάρχουν και κάποια θέματα ε, με τα οποία δεν ταυτιζόμαστε. Τα ε, περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα που ε, ε, τα αναφέρει ως ε, συντονιστικά κέντρα. Ε, καταρχάς να συγχαρώ τον εισηγητή για το ότι βρήκε το σωστό όρο. Αυτό θέλαμε να πούμε κι εμείς. Λέγοντας ε, cooperation, ε, coordination centers. Δεν θέλαμε στην πραγματικότητα να δημιουργήσουμε νέες δομές. Ποτέ, ποτέ δεν ήταν σκοπός μας να δημιουργήσουμε νέες δομές ε, που θα δυσκολεύουν το έργο. Αντίθετα, ο όρος του εισηγητή είναι εξαιρετικός και ακριβώς αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Δεύτερο θέμα. Τα καθήκοντα. Εδώ κάναμε μια πρόταση η οποία, με την οποία συμφωνεί σε μεγάλο βαθμό και ο εισηγητής. Ακούσαμε για τα στοιχεία ετοιμότητας έναντι των κινδύνων που ε, διαγράφονται από την έκθεση. Εγώ τοποθετήθηκα ήδη για αυτό το θέμα και υπάρχει και το ζήτημα της αρμοδιότητας λήψης αποφάσεων. Εδώ, σε αυτό το στον τομέα, αυτό που βλέπω στην έκθεση μου προκαλεί σύγχυση, ως νομικού πρέπει να σας πω, διότι υπάρχει μια διάκριση μεταξύ της σύστασης, όπου τα κράτη-μέλη έχουν τη δυνατότητα βεβαίως να αποκλείουν και υπάρχουν και οι κανονικές ε, συστάσεις. Δεν καταλαβαίνω όμως ποια ακριβώς είναι η διαφορά μεταξύ των δύο ενιών. Θα ήθελα λοιπόν να καλέσω τον ε, εισηγητή να ξανασευτεί το θέμα. Στις δύο λειτουργίες που υπάρχουν συστάσεις με δυνατότητα απόκλησης, ίσως δεν θα έπρεπε σε αυτή την, σε αυτή περίπτωση να αποκαλούνται ως αποφάσεις με δυνατότητα απόκλησης για λόγους ασφαλείας και όλα τα άλλα να είναι συστάσεις που δεν θα είναι νομικά δεσμευτικές. Πολύ σύντομα για την ε, τροφοδότηση κατά προτεραιότητα των ανανεώσιμων. Εγώ συμφωνώ με όσα είπαν ο κύριος, η κυρία Βέρνερ, ο κύριος Τούρμες. Νομίζω ότι εδώ η Κομισιόν κατάφερε να ε, επιτύχει σωστή ισορροπία. Αντιθέτως νομίζω ότι ο εισηγητής ίσως υπερβαίνει κάπως τα, τα όρια αυτή τη στιγμή. Και ισχύει αυτό που είπε ο κύριος ε, Τούρμες με δεδομένο ότι δεν υπάρχει ακόμα μια πλήρως εύρυθμη και ε, ε ενιαία αγορά, ε, δεν γίνεται να προχωρήσουμε υπερβολικά, ε, σε υπερβολικά μεγάλο βάθος. Εγώ πιστεύω ότι η φόρμουλα που βρήκατε για το DSO είναι ακριβώς σωστή. Γιατί να υπάρχει διαφορά στον, στον ορισμό. Ε, όσο προς τις υποχρεώσεις TSO και DSO, γιατί εκεί αναφέρεται ότι τα αποθέματα περιορίζονται πραγματικά ε, ε, σε κάτι που δεν μπορεί να παράσχει η αγορά. Ενώ η TSO είναι πάρα πολύ ευρύς όρος, καθώς είναι οποιοδήποτε εμπλέκεται στο σύστημα μεταφοράς. Γι' αυτό χωράει πολύ ευρεία ερμηνεία. Για την έκθεση για την οδηγία, εδώ χαιρετίζουμε τις προσπάθειες που έχει καταβάλει ο εισηγητής προκειμένου να αυξηθεί το επίπεδο προστασίας των καταναλωτών, την αλλαγή από πάροχο σε πάροχο. Το 2025 θεωρώ ότι είναι πολύ καλή προθεσμία, ανεξαρτησία των συγκριτικών εργαλείων, αποσαφήνιση των ε, όρων και των πληροφοριών της τιμολόγησης, όλα αυτά, με όλα αυτά συμφωνούμε. Για τις ρυθμισμένες τιμές. Εδώ θα ήθελα να ε, επιστήσω την προσοχή σας. Από την εμπειρία μου, όταν προσπαθήσαμε ως Γενική Διεύθυνση να πείσουμε τα κράτη-μέλη να απαλλαγούν από τις ρυθμισμένες τιμές και να εισάγουν ένα νέο σύστημα, τι κάναμε. Πρώτον, δημιουργήσαμε ένα ε, στεναρό σύστημα για την προστασία των, ε, των ευάλωτων καταναλωτών. Προτού προχωρήσουμε στην απελευθέρωση. Για να το κάνεις αυτό όμως χρειάζεσαι ε, μια μεταβατική περίοδο και ορισμένους κοινωνικούς δείκτες. Γιατί δεν μπορείς εν μία νυχτή να δημιουργήσεις μια κοινωνική πολιτική ε, μάλλον μέσω της κοινωνικής πολιτικής, όλα τα απαραίτητα εργαλεία και τα συστήματα. Γι' αυτό και σε αυτές τις περιπτώσεις πάντοτε είναι πάντοτε χρήσιμο, χρήσιμο να υπάρχουν μεταβατικές περίοδοι. Να, υπάρχουν δηλαδή, να υπάρχει κάποια μεταβατική περίοδος με συγκεκριμένους κοινωνικούς δείκτες και από εκεί και πέρα, αφού ολοκληρωθεί αυτή η μεταβατική περίοδος, να περάσει στην πλήρη απελευθέρωση. Ο κύριος Τούρμες είπε ότι δεν πρέπει να ρυθμίζονται οι τιμές, αλλά τα περιθώρια. Το κάνουν κάποια κράτη-μέλη. Ωστόσο, πώς τότε δίνουμε τα σωστά σήματα για επενδύσεις αν ρυθμίζονται τα περιθώρια κέρδους ε, στην, στην αγορά. Γιατί πρέπει με την πρότασή μας να ε, δώσουμε και τα σωστά, να στείλουμε και τα σωστά μηνύματα στο, στους επενδυτές. Για την αποζημίωση ε, υπάρχει το ζήτημα. Ναι, ή όχι. Αυτό που επιλέξαμε εμεί να κάνουμε είναι ότι δεν θα υπάρχει αποζημίωση, αλλά η Εθνική διευθυντική Αρχή μπορεί, εφόσον υπάρχουν λόγοι, να προβλέπει ε, κάτι τέτοιο. Τώρα ο εισηγητή το αντιστρέφει αυτό και λέει αποζημίωση εκτός αν υπάρχουν λόγοι για να μην καταβλεί αποζημίωση. Εμείς λοιπόν ε, καταλήξαμε στο, στη μη αποζημίωση ως αρχή, διότι αν το αντιστρέψει κανείς, όπως γίνεται στην έκθεση, υπάρχει, ε, ε, αποτελεί κάτι τέτοιο εμπόδιο για τους aggregators, για την είσοδό τους στην αγορά. Και αυτό δεν θα μας βοηθήσει στο να ε, κατακτήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα είναι ανοιχτό και αξιόπιστο και θα προσελκύει όσο το δυνατόν περισσότερους παίκτες. Αυτά συνολικά πάντως να σας πω ότι έχουν κατατεθεί πάρα πολλές ε, και πολύ ενδιαφέρουσες ε, ε, προτάσεις και στις δύο εκθέσεις. Η Κομισιόν πράγματι, πραγματικά χαιρετίζει την συνολική δομή αλλά και την προσέγγιση που επέλεξε ο εισηγητής αλλά και που από ό,τι άκουσα σήμερα την χάνει και της ευρύτατης συμφωνίας από τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής σας. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Κύριε Κρισιάνης. Να σας πω πως είναι εξαιρετική η εκθέσή σας, το είπαν και οι συνάδελφοι αγαπητέ Κρυσάνης, αλλά πολλά πρέπει να αλλάξει. Σας αυτή την εξαιρετική έκθεση, επαναλαμβάνω. Όλοι σας έδωσαν συγχαρητήρια και όλοι είπαν ότι ήταν πολύ καλή έκθεση. Τώρα αλλαγές. Πώς σου φαίνεται. Εξαιρετικά σχόλια θα απαντούσα εγώ. Αλλά ε, όταν ακούω τα όσα λένε οι συνάδελφοι, κάποιες από τις προτάσεις για τη βελτίωση νομίζω ότι είναι αντικρουόμενες. Και το πρώτο το οποίο χρειάζεται να αποφασίσουμε και το οποίο πρέπει να δούμε σε όλες τις πολιτικές ομάδες είναι θέλουμε να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε την κατεύθυνση στην οποία ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δηλαδή να μπει η έννοια της αγοράς στην κατάσταση της ηλεκτρικής ενέργειας. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή αγορά για την ηλεκτρική ε, αγορά. Έχουμε μια πολύ κατακαιρισματισμένη αγορά με πολύ διαφορετικές καταστάσεις επιτόπου. Άλλο η Ισπανία που έχει τεράστιο δυναμικό σε ΑΠΕ αλλά δεν έχει τη δυνατότητα εξαγωγής Η Γαλλία έχει ένα σύστημα το οποίο ανέπτυξε πριν από 30-40 χρόνια το οποίο βασίζεται στην πυρηνική ενέργεια και το οποίο δεν είναι και πολύ ευέλικτο. Οπότε ίσως αυτοί οι οποίοι δεν είναι ευέλικτοι δεν θέλουν να επιτρέψουν να μπει η ευελιξία γιατί ξέρετε ότι ώρες μέσα στην ημέρα θα είναι πάμφθινη η ενέργεια ηλιακή από την ε, η φωτοβολταϊκή από την Ισπανία, οπότε κάποιοι μπορεί να μην θέλουν αυτές τις χαμηλές τιμές να μπαίνουν στη Γαλλία. Και στη Γερμανία, να σας πω, δεν υπάρχουν αρκετές γραμμές μεταξύ του βορρά που παράγει πολλά, πολλή ενέργεια και του νότου που στη Γερμανία καταναλώνει πάρα πολύ ενέργεια. Δεν ξέρω είναι κάποιες ε, ε, κοινότητες που δεν ε, θέλουν να έχουν αυτές τις γραμμές υψηλές τάσεις στο ε, περιβάλλον τους, αλλά εν πάση η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι εύκολη σαν το φυσικό αέριο να αποθυματοποιηθεί και πολλές φορές δεν μπορεί να πάει εκεί που τους στέλνουμε. Οπότε πολλές φορές έχουν ακολουθήσει την τακτική της ίσονος αντίστασης και αυτό έχει οδηγήσει στο να πηγαίνουμε από τη Τσεχία στην Αυστρία και Τούμπαλη και από εκεί στο νότο της Γερμανίας Όλα αυτά αποτελούν την πραγματικότητα και δημιουργούν πρόβλημα για τις χώρες που ε, προσπαθούν να στείλουν αυτή την ενέργεια. Η Πολωνία είναι διαφορετική, λίγο παρόμοια με τη Γερμανία. Έχει μεγάλο στόλο μη ε, ε, ευέλικτης παραγωγής, άνθρακα, όχι πυρηνική, αλλά και εκεί υπάρχουν κάποιες ιδιάζουσες συνθήκες. Οπότε αυτό που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είναι σωστό είναι ότι δείχνει μια κατεύθυνση και λέει προ τα εκεί θέλουμε να πάμε. Και εμεί θα πρέπει ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δούμε. Θέλουμε να αποφασίσουμε ότι αυτή είναι η κατεύθυνση. Δεν θα το καταφέρουμε σε μια μέρα. Αυτέ είναι επενδύσει που πρέπει να γίνουν σε 20-30 χρόνια. Δεν θα γίνει εν μία νυχτή, αλλά για του επενδυτέ είναι καλό να γνωρίζουν ποια είναι η κατεύθυνση προ την οποία στοχεύουμε. Μηχανισμοί δυναμικότητα. Ούτε με να μ' αρέσουν οι επιδοτήσει ε, για το πυρηνικό, όπως δεν μου αρέσουν και οι επιδοτήσεις για τις ΑΠΕ. Προσπάθησα να το κάνω ξεκάθαρο και σε πνευματικό επίπεδο φεύγουμε από εκεί και πάμε προς την ε, τακτική της αγοράς που δεν επιδοτούμε. Αλλά πουθενά δεν μιλώ για αναδρομικές αλλαγές. Μία πρόταση να κοιτάξουν τα κράτη-μέλη, αν υπάρχει τρόπος, θα το πω, ανοιχτά, να εξαγοράσουν τις υφιστάμενες συμβάσει. έτσι ώστε να μην πληρώνουν για 10-15 χρόνια στο μέλλον, ελάτε να τους εξαγοράσετε σήμερα. Και σε ένα κράτο μέλος αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σε άλλο όχι. Πάντως είναι η γενικότερη κατεύθυνση, θα δούμε όλα τα σημαντικά και το priority dispatch και τα λοιπά, δηλαδή την καταπροτεραιότητα αποστολή, αλλά πρέπει να δούμε τι γίνεται για τα 550, βέβαια, αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα για τις περιοχές της Ευρώπης που έχουν πολλούς που ε, δουλεύουν σε ανθρακοριχεία. Μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά πρέπει να το δούμε. Και για την ενεργειακή ένδια, και εκεί υπάρχουν δύο διαφορετικές προσεγγίσεις. Είτε επιδότηση τιμών, έτσι ώστε να μειωθούν οι τιμές, είτε επιδότηση ε, Και εγώ πάντα λέω ότι καλό είναι να μην στρεβλώνει κανείς τις αγορές με ρύθμιση ε, στην αγορά, αλλά να επιδοτεί κανείς κάποιους να μπορούν να πληρώσουν τους λογαριασμούς τους. Αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος. Δηλαδή, όσο το δυνατόν λιγότερη στρέβλωση και με χαρά θα συνεργαστώ με όλους σας, θα τα καταφέρουμε. Thank you very much, Christianis, for your... Ευχαριστώ, Κριστιανής, για όλη τη δουλειά που έχεις κάνει. Έχουμε μία παγκόσμια αγορά για το αργό, για το φυσικό αέριο, αλλά χρειάζεται και μία ευρωπαϊκή ενεργειακή αγορά. Ευχαριστώ πολύ. Προθεσμίες. 15 Σεπτεμβρίου. 15 Σεπτεμβρίου προθεσμία για τις τροπολογίες. Και το απόγευμα η συνάντησή μας θα γίνει στο 6Q1, όχι εδώ μέσα, εκεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Και ευχαριστώ τους που όλοι είχαμε την τύχη, 12.30 ακριβώς, να κλείσουμε τις συνεδρία. Ευχαριστώ πολύ.